Gentlemen, Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε. Έχουμε άφθονα σημεία στην ημερήσια διάταξη. Επειδή δεν μπορέσαμε να συναντηθούμε τη Δευτέρα, παρακαλώ τώρα ησυχάστε. Please, please, please. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ πολύ συνάδελφοι. Thank you. Ε- Ευχαριστώ. Επειδή τη Δευτέρα δεν μπορέσαμε να συνεδριάσουμε και παρόλα αυτά έπρεπε κάποιες αποφάσεις να ληφθούν για κάποια σημεία της Δευτέρας, ε, κάποια τα κράτησα λοιπόν και τα έχω μεταφέρει στη σημερινή συνεδρίαση. Πρέπει λοιπόν να είμαστε γοργοί στην εξέταση των θεμάτων για να καλύψουμε αυτή την εκτεταμένη μερίσια διάταξη. Έχουμε λοιπόν την περασμένη μερίσια διάταξη συν καθώς και τα σημεία 6, 7, 11 και 5 τα οποία μετακινήθηκαν από την ημερήσια διάταξη της Δευτέρας. Έχουμε όμως και άλλα σημεία και λίγο χρόνο πρέπει να βιαστούμε. Αντιρρήσεις για την ημερήσια διάταξη. Αλλαγές πέραν αυτών που σας ανακοίνωσα. Ωραία λοιπόν. Έγκριση πρακτικών της συνεδρίασης 21 Αυγούστου. Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις στο τέλος αυτής της συνεδρίασης, θεωρούνται εγκεκριμένα. Αλλαγή στα πρακτικά. Διότι εφ' εξής, τα πρακτικά θα περιλαμβάνουν σύνοψη των αποφάσεων και συστάσεων που ε, λαμβάνονται στην συνεδρία των συντονιστών στις ίδιες ημερομηνίες για σκοπούς διαφάνειας, διότι υπήρξαν παράπονα για την έλλειψη ενημέρωση του κοινού για τις αποφάσεις μας στις συναντήσει των συντονιστών. Δεν θα υπάρξει λοιπόν καταγραφή των συζητήσεων των συντονιστών, αλλά των αποφάσεων και συστάσεων τους. Uh Um, Έχετε στα έδρανά σας τα φυλάδια της, συνάντηση. της συνάντησης. της 21ης και 22ης Αυγούστου και πριν την διακοπή της 19ης Σεπτεμβρίου. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Έχουμε web streaming ως συνήθως. Όπως σας ενημέρωσα, Επειδή δεν έγινε συνάντηση της Δευτέρας, έπρεπε να επιλέξω ποια θέματα μπορούμε να δούμε σήμερα. Αυτά που ήταν πιο επίγοντα και στα οποία έπρεπε να ληφθεί απόφαση λόγω χρονοδιαγράμματος. Δύο λοιπόν σημεία, Ουσμπεκιστάν και Ισραήλ, με τις σχετικές συμφωνίες, αυτά θα τα δούμε στις 11 Οκτωβρίου τότε θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών για το θέμα του Ουσμπεκιστάν, την έκθεση του Ουσμπεκιστάν, ήταν 22 Σεπτεμβρίου, αλλά παρατείνεται στις 14 Οκτωβρίου. Επαναλαμβάνω, τροπολογίες για την έκθεση του Ουσμπεκιστάν 14 Οκτωβρίου το μεσημέρι στις 12 η ώρα. Και τα δύο θέματα, το Ουσμπεκιστάν και το Ισραήλ, θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διατάξη τη συνάντησης τη 11 η Οκτωβρίου. Calendar. is... Το χρονοδιάγραμμα από το πρόγραμμα της Δευτέρας πλοβρέπει την ε, απόφαση που ελήφθη 21 Αυγούστου από τους συντονιστές ε, μετά εγκρίθηκε και από την Επιτροπή, οπότε αν δεν υπάρχει αντίρρηση το χρονοδιάγραμμά μας παραμένει ως εγκρίθηκε. Adopted. Item 6. Σημείο 6. Κατάσταση του τριμερούς διαλόγου. Πληροφόρηση από τους εισηγητές για τις συμφωνίες διμερών επενδύσεων. Μετά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια, οι συντονιστέ μα το συζήτησαν. Υπήρξε δεύτερο γύρο τριμερού διαλόγου. Προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιες, ε, κάποια σημεία συμφωνία για τι αντιφάσει που υπήρχαν μεταξύ Συμβουλίου και ημών και η Επιτροπή προσπάθησε να κατανοήσει καλύτερα τη δική μας τάση. Έπειτα ζητήθηκε από την Επιτροπή να προετοιμάσει τις μελλοντικέ συζητήσεις όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτά είναι, αυτές είναι οι εξελίξεις σε σχέση με το θέμα. Έκθεση για το ICI. συμμετείχαμε στη συνδιαλλαγή με το Συμβούλιο, επιτελέστη πρόοδος, ακολουθήσαμε μία ενιαία μέθοδο, δεν θα συμφωνείτε τίποτα μέχρι όλα να έχουν συμφωνηθεί. Το θέμα του ICI έχει φτάσει στο σημείο του συμβιβασμού Εάν λοιπόν συμφωνήσουμε και στο άλλο σκέλος, θα υπάρξει τελική συμφωνία και για τα δύο. Μέχρι να γίνει αυτό, δεν θεωρείται συμφωνηθέν το θέμα. Όμως, οι συζητήσεις για το ICI πήγαν καλά και εκφράζω την ικανοποίησή μου. Ε, με τη βοήθεια του συναδέλφου και με τη δική μου τη συνδρομή και με τη στήριξη των ε, πολιτικών ομάδων πετύχαμε το επιθό αποτέλεσμα. Ε, έκθεση για κολλήνο. Υπήρξαν και κάποιες ε, αντιφάσεις μεταξύ των απόψεων του Συμβουλίου και της δικής μας. Και κάποιες φορές λόγω παραπληροφόρησης απλώς. Έγινε λοιπόν μια άτυπη συνάντηση και επετέχθη συμφωνία. Ζαντό, έκθεση Ζαντό για τις ψαγωγικές ε, πιστώσεις. Συμφωνία το Σεπτέμβριο και πιστεύουμε ότι η συμφωνία μας θα βελτιώσει το βαθμό διαφάνειας που διέπει αυτό το θέμα. Έχει έρθει ο κύριος Ζαντό. Ίσως να θέλει κάτι να μας πει για τις εκθέσεις αυτές. Κάποιος να μιλήσει για την έκθεση ICI, για τη συνδιαλλαγή. The Πρόοδος στο θέμα αυτό. Εγώ ήδη είπα στους συναδέλφους τη δική μου την οπτική την άποψη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μόλις έφτασα γιατί είχα κολλήσει στη συμφόρηση την κυκλοφοριακή λόγω της διαδήλωσης στη Λουά. Σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι ως διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου όλα τα μέλη πιστεύουμε ότι χρειάζεται κοινή λύση για όλα τα μέσα. Θέλουμε να βρεθούν συμμεβαστικές λύσεις όσο το δυνατόν περισσότερε στον συνεχιζόμενο τριμερή διάλογο για το χρηματοδοτικό μέσο για το ici αυτό σημαίνει ότι η κοινή μας λύση πρέπει να διασφαλίζει και να εγγυάται ότι το Κοινοβούλιο θα έχει δικαίωμα λόγου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα οικονομικά αυτά μέσα, τα οικονομικά εργαλεία για τις πολιτικές μας. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να διατηρήσουμε την ισορροπία και την συνεπή προσέγγιση του Ευρωκοινοβουλίου και σε επίπεδο Επιτροπή ΣΥΝΤΑ και σε συνεργασία με τι υπόλοιπε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ που συνεργάζονται σε αυτόν τον τριμερή διάλογο. Θα γίνει τίποτα στο Στρασβούργο. Ο τελικός γύρος ίσως. Κοίτα ίσως για να πετύχουμε την ε, τελική συμφωνία. αν πετύχουμε συμφωνία λοιπόν στον ΦΑΚΕΡ στο θέμα ICI ε, και στο άλλο, παρόλο που υπήρχαν, ε, ήταν αμφιλεγόμενο, θα είναι μια επιτυχία. Ο κύριος Ζικολίνο είναι εδώ. Τίποτα να μας πείτε και εσείς για τη δική σας έκθεση για το πρωτόκολλο ΦΥΡΟΜ. Έχει κλείσει και αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, με συγχωρείτε για την καθυστέρηση που σημείωσα. Όπως σωστά είπατε λίγο πριν, τα πράγματα πάνε αρκετά καλά. Έχει κλείσει οριστικά ο τριμερής διάλογος με τις μικρές γλωσσικές ατέλειες που απομένουν, τις οποίες όμως ξεπεράσαμε εν μέρη. Πιστεύω ότι ο ορισμός που στον οποίο καταλήξαμε είναι σκόπιμη λύση. Ο τριμερής διάλογος σύντομα, χάρη στη συμβολή του, Συμβουλίου, κατάφερε αυτό το αποτέλεσμα. Και βεβαίως χάρη στη στήριξη των σκιωδών εισηγητών. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Από τους τέσσερις λοιπόν φακέλους, σε δύο έχουμε επιτυχές αποτέλεσμα. Και στον ένα έχουμε σχεδόν τελικό αποτέλεσμα και συμφωνία. Ενώ οι συμφωνίε διμερών επενδύσεων, ή μάλλον διμερεί συμφωνίε επενδύσεων, βρίσκονται στην αρχή των συζητήσεων. Θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί λύση. Περνάμε στο σημείο 7. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ακριβώς για τα ζητήματα που ανέφερα. Έκθεση Σαλβατόρε Γιακολίνο. για το πρωτόκολλο των πυροβολών όπλων. Vote on the agreed compromise Ψηφοφορία για το κείμενο της, ε, όπως τροποποιήθηκε. Μία ενιαία ψηφοφορία. Ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Sorry. My card is not okay. Correctly inserted. It is already. The vote is. I have 19 people there and only 18 votes. Πέρας, 21 είναι παρόντες, 18 ψήφισαν. Πέρας της προφορίας λοιπόν. Εγκρίθηκε ομόφωνα. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, τον κύριο Γιακολίνο. Και τώρα ψηφίζουμε την έκθεση του Νικολό Ρινάλντι για την κατάσταση υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Κεντρική Ασία. Έχουμε περίπου 40 τροπολογίες είναι γνωμοδότηση της τα καθήλυνα αρμόδια επιτροπής. Ας περάσουμε στην ψηφοφορία. Υπάρχουν κάποιες συμβεβαστικές τροπολογίες. Οπότε μειώνεται ο συνολικός αριθμός τροπολογιών.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 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 17 και 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 20. Is open. Amendment. Άρχεται η ψηφοφορία. 20. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίφθηκε. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 λέει ο πρόεδρο. 34 διορθώνει. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική. Άρχεται. And the vote is closed. Και λίγη πέρας. Εγκρίθηκε με 17 ψήφους υπέρ και 4 κατά. Συγχαρητήρια στον κύριο Ρινάλντι. This uh, Φτάσαμε στο τέλος των ψηφοφοριών. Προχωρούμε στο σημείο 9, φραγμή στο εμπόριο και τις επενδύσεις. Έκθεση πρωτοβουλίας δική μας. Ο Ρόμπερτ Στέρντι είναι ο εισηγητής. μετά την ανακοίνωση της Κομισιόν για τους φραγμούς του εμπόριο και τις επενδύσεις το 2011 και δίνω το λόγο στον εισηγητή που είναι εδώ, ο κύριος Ρόμπερτ Στέρντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η έκθεση πρωτοβουλίας γιατί γνωρίζετε καλά και το είπε και ο Πρόεδρος τώρα το Φεβρουάριο φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση για τους φραγμούς στο εμπόριο και την, ε, τις επενδύσεις ε, και ζητεί να βελτιώσουν την πρόσβαση στην αγορά οι οικονομικοί εταίροι, να καταργήσουν ε, τους φραγμούς στο εμπόριο και επίσης θα επανεξετάσει το θέμα αυτό το Μάρτιο του χρόνου. Γι' αυτό λοιπόν, αν προλάβουμε να περάσουμε την έκθεση από την Ολομέλεια μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, πριν από τα Χριστούγεννα δηλαδή, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί θα ενισχύσει τη θέση μας σε σχέση με την Κομισιόν. Η ίδια η έκθεση ε, παρουσιάζει εκτενή επισκόπηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω μη δασμολογικών εμποδίων. Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα των εμποδίων. Μιλάμε με τις επιχειρήσεις στις πατρίδες μας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακολουθήσαμε και τις εμπορικές διαπραγματεύσεις εδώ στις Βρυξέλλες. Ε, παρά τις προσπάθειες ελευθέρωσης, ε, περιοριστήκαμε στην κατάργηση των δασμών. Αλλά δαπανηρά, τα δαπανηρά αυτά εμπόδια ε, γίνονται πιο ανησυχητικά. Υπάρχουν ε, ενδείξεις που δείχνουν ότι οι χώρες προσφεύγουν όλο και περισσότερο σε αυτά τα προστατευτικά μέτρα. Αν δούμε την Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με την Κορέα που ήταν η πρώτη που απασχόλησε το Κοινοβούλιο, αρχίσαμε να βλέπουμε τι γίνεται όταν βλέπαμε τους εισηγητές ακόμα και στους μηχανισμούς διασφάλισης και τις συμφωνίες τις εμπορικές που προσεγγίζονταν από μέλη διαφόρων λόμπι συνεχώς και εμείς για ε, το διεθνές εμπόριο και τους φραγμούς εκεί. Είναι σημαντικό λοιπόν να προχωρήσουμε πέρα από τα προβλήματα που εντόπισε η Κομισιόν, να δούμε και εμείς ε, τα ίδια, δεν θα ήταν επικοδομητικό. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τις καταχρήσεις χωρίς προκαταλήψεις και να δούμε τη ρίζα του κακού. Υπάρχουν πολλά θέματα αυτό που προσπάθησα να κάνω στην έκθεση είναι όχι να την ε, φορτώσω από διάφορους εμπορικούς φραγμούς που μας ε, κοινοποιούν, γιατί θα υπάρχει δυνατότητα και μέσα από τις τροπολογίες να καταδειχθούν αυτά τα φαινόμενα. Α, μπορούμε να καταγράψουμε χιλιάδες τέτοιες εμπορικές συμφωνίες ε, με όλους και έτσι κι ε, είναι περιορισμένε οι εκθέσει που μπορούμε να υποβάλουμε. Στο δεύτερο μισό λοιπόν του κειμένου προσπαθώ να κάνω κάποιες απλές αλλά ξεκάθαρες συστάσεις για αποφασιστικές ε, δράσεις ε, από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Ελπίζω η Κομισιόν να εξετάσει τις συστάσεις σε σχέση με την έκθεση του 2012 και μέσω μακροπρόθεσμα να εφαρμόσει τις συστάσεις αυτές. Γι' αυτό πρέπει να προλάβουμε να περάσει από το Κοινοβούλιο και να φτάσει στην Κομισιόν τέλος του χρόνου η έκθεση αυτή. Και κάτι, ένα άλλο πρόβλημα που δεν είναι εμπορικός φραγμός και εμπόδιο, το συζητήσαμε στους συντονιστές όταν συζητάγαμε για τις προτάσεις Ομπάμα, δεν είναι διεθνές ε, εμπορικό εμπόδιο, αλλά αρχίζομαι να βλέπουμε αυτό το ρεφλέξ. Αν δεν προσέξουμε, ε, ο προστατευτισμός περνάει μέσα από τέτοιου είδους ε, μέτρα και εμπόδια και κάτω από δύσκολες συνθήκες ε, προσπαθεί ο καθένας να βοηθήσει τη χώρα του σηκώνοντα εμπορικά εμπόδια και φραγμούς και αυτό θεωρώ ότι καταστρέφει τις ευκαιρίες που έχουμε για να βγούμε από τις χρηματοπιστωτικές μας δυσκολίες. Και τώρα περιμένω με ενδιαφέρον κύριε Πρόεδρε να δω τι θα πούν οι συναδέλφοι. Ευχαριστώ πολύ. Σκιώδης. Φιάλνερ από το ΕΛΚ. Έχεις πολύ, Ρόμπερτ, για την εισαγωγή. Όπως είπατε, είναι σημαντικό θέμα και νομίζω ότι η έκθεσή σας είναι καλή. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι δασμοί δεν είναι αυτό που απασχολεί πιο πολύ τους επιχειρηματίες, την επιχειρηματική κοινότητα. Υπάρχει και αυτό το θέμα, αλλά κυρίως, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι οι μη δασμολογικοί ε, φραγμοί που τους απασχολούν. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε την εμπειρία που υπάρχει όταν μιλάμε για μη δασμολογικούς φραγμούς την εμπειρία της Ένωσης, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση χτίστηκε πάνω στην ιδέα της δημιουργίας ενιαίας αγοράς με κατάργηση των εμπορικών φραγμών στους κόλπους της Ένωσης. Πολλά διδάγματα μπορούν να αντληθούν λοιπόν από τα 57 χρόνια τέτοιων προσπαθειών στην Ευρώπη και πώς μπορεί αυτό το σύστημα να επεκταθεί σε όλο τον κόσμο. Ε, ίσως δεν θα είμαι, θα είμαι κάπως αντισυμβατικός, θα επανέλθω μέσα από τροπολογίες για να πω ότι κάτι το οποίο έχουμε ξεκαθαρίσει αρκετά καλά είναι να δημιουργήσουμε ένα μέσο το οποίο καταργεί κάποιους φραγμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν το θέλει όμως κανείς στην πραγματικότητα. Έχουμε μη δασμολογικούς φραγμούς και για προστατευτικούς λόγους από διάφορες χώρες, αλλά πολλές φορές πρόκειται για έλλειψη συνεργασίας, διαφορετικά πρότυπα, Δηλαδή είναι τυχαίοι κάπως, αν θέλετε, ε, μη σκόπιμη, μη δασμολογική φραγμή. Και στην Ευρώπη εμείς ε, έχουμε το Solvit στην ε, εσωτερική αγορά, ε, τον οργανισμό που πρέπει να έχει κάθε κράτος μέλος και θα πρέπει εκεί να αναφέρονται οι επιχειρήσεις αν απαντούν δυσκολίες στην εσωτερική αγορά και φραγμούς. Υπάρχουν πολλά στοιχεία, νούμερα, συμβουλές και υπάρχει και παροχή βοήθειας για να καταργηθούν οι φραγμοί. Πολλές φορές λέω γιατί να μην λειτουργεί και αυτό στον ΠΟΕ, ο ΠΟΕ δηλαδή γιατί να μην βοηθάει καταγράφοντας αφενός κατά περίπτωση τα περιστατικά αυτά, αντλώντας από την επιτυχή εμπειρία της Ευρώπης μέσα από το Solvit, αν και θα ήταν κάπως αντισυμβατικό, ε, νομίζω ότι θα ήταν τουλάχιστον μια ιδέα που μπορούμε να προωθήσουμε, να αξιοποιήσουμε δηλαδή την εμπειρία από το Solvit για να καταπιαστούμε με παγκόσμια προβλήματα σε μη δασμολογικού φραγμούς. Υπάρχουν βέβαια και τομεί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έκανε αρκετά μεν, αλλά καλύτερα είμαστε εμείς από ό,τι είναι η κατάσταση παγκοσμίω. Και τώρα το πιο σημαντικό για τους οικονομικούς επιχειρηματίες και τους παράγοντες είναι το η παγκόσμια αρένα. Ε, θα ήθελα στην έκθεσή σας να αναφερθεί πιο πολύ το θέμα των υπηρεσιών, εμπόριο των υπηρεσιών. Αυξανόμενος ο όγκος τους, το πιο σημαντικό κομμάτι του παγκοσμίου εμπορίου είναι οι υπηρεσίες σήμερα και έχουμε τεράστιους εμπαρικούς φραγμούς στον τομέα των υπηρεσιών. Γι' αυτό λοιπόν θα ε, καταθέσω τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση ούτως ώστε να ενισχύσω τα επιχειρήματά μας για το πώς θα μπορέσουμε να καταργήσουμε τους μη εμπορικούς ε, φραγμούς και τους ε, εμπορικούς φραγμούς στις ε, υπηρεσίες. Ψηφιακή οικονομία. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Δεν έχει σύνορα το διαδίκτυο σήμερα, αλλά δυστυχώς πολύ εμπόριο στην ψηφιακή οικονομία μέσα από το διαδίκτυο εμποδίζεται από τα σύνορα. Η διαδικτυακή οικονομία δεν πρέπει να έχει τέτοια εμπόδια. Δεν είναι φυσικό αυτό το πράγμα, είναι αφύσικο. Ε, υπάρχουν λοιπόν και εδώ εμπόδια. Τρία πράγματα λοιπόν θα με απασχολήσουν στις τροπολογίες μου. Πρώτον, θα προσθέσω κάποιες ιδέες για το πώς θα μπορέσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο να μάθουμε από την εμπειρία του Solvit. Δεύτερον, ε, θα τονίσω τις υπηρεσίες και τους φραγμούς που υπάρχουν εκεί στις υπηρεσίες. Και τέλος, πολύ σημαντικό, η ψηφιακή οικονομία και πώς θα ε, καταργήσουμε παγκοσμίω τους φραγμούς στην ψηφιακή οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Επόμενος Κιώδης. Καταρρίφ, δεν μπορούσε όμως να έρθει, γιατί έχασε την πτήση προς Βρυξέλλες. Μου ζήτησε όμως να διαβάσω τα σχόλιά του. Proxy, SND, Shadow. Ε, Θα σας τα διαβάσω λοιπόν για το, το θέμα αυτό. Είναι στα γαλλικά. Θα σας τα διαβάσω όσοι έχουν, λέει ο πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Στέρντι για το σχέδιο έκθεσής του. Ακόμα και αν λυπάμαι που η δικιά μας Επιτροπή δεν μπόρεσε να έχει ανταλλαγή απόψεων προηγουμένως ε, για αυτό το τόσο ουσιαστικό θέμα εξετάζοντας σε βάθος την πρόταση της Επιτροπής, θα μας βοηθούσε να προχωρήσουμε σε μια τέτοια μακροχρόνια δουλειά και σήμερα βρισκόμαστε υποπίεση, μια που η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών θα είναι αύριο. Ήθελα λοιπόν να εκφράσω τη διαφωνία μου για τη διαδικασία αυτή. Επί της ουσίας τώρα, η έκθεση του κυρίου Στέρντι τα βάζει με πραγματικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις αγορές ορισμένων τρίτων χωρών. Μιλάει για την καταπολέμηση μασκαρεμένων μέτρων που δυσκολεύουν την πρόσβαση στην αγορά των επιχειρήσεών μας, ενώ η ευρωπαϊκή αγορά είναι ανοιχτή και υποβάλλεται στον ανταγωνισμό απ' έξω. Ένα τέτοιο άνοιγμα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για στοιχεία τα οποία και εγώ ίδιο έχω αναπτύξει στη γνωμοδότηση που ετοίμασα εγώ για τι δημόσιε αγορέ και από εκεί θα εμπνευστώ για να προσπαθήσω να συμπληρώσω την έκθεση, κατά τα άλλα ξέρετε, του κύριου Στάρντι. Χαίρομαι για την έκθεση αυτή και βλέπω και εγώ ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία και διάλογος έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τους μη δασμολογικούς περιορισμούς. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιοι μη δασμολογικοί φραγμοί, γιατί αν τους αφήσουμε, αυτό θα ήταν λάθος και σε βάρος του εμπορίου μας. Τέτοια μέτρα δεν είναι καν προστατευτικά. Είναι μέτρα πολλές φορές που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία ή που έχουν να κάνουν με ειδικά αιτήματα των πολιτών. Και για παράδειγμα θα σας αναφέρω το εξής. Η ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά την ε, άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δεχτεί γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ή βόλιο κρέας με ορμόνες, αυτά τα πράγματα είναι πολιτικές που ορισμένοι δικοί μας ε, ε, εταίροι θεωρούν ότι είναι μη δασμολογική φραγμή. Όμως δεν είναι έτσι, γιατί αυτά έχουν να κάνουν με την δημόσια υγεία και πρέπει να υπάρχουν. Ε, προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θα προσπαθήσω να ενισχύσω την έκθεση Στέρντι με τροπολογίες τις οποίες ελπίζω να υποστηρίξουν οι περισσότεροι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ. Η θέση των ε, σοσιαλιστών λοιπόν συμπληρώνεται ως εξής. Η κυρία Μουσκαρντίνη έχει το λόγο. Ήταν ε, πολύ ενδελεχής η όλη προσπάθεια, χάρη στη συνδρομή και των υπολείπων συναδέλφων και γι' αυτό ήταν πλήρης η εξέταση του θέματος. Απλώς, παίρνοντας αφορμή από όσα είπε ο κ. Χέλνε προηγουμένως και από τα σχόλια που έκανε ο Ρόμπερτ με την παρουσίαση που μας διαβάσατε για τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Θα συμμετάσχουμε ως Επιτροπή και στη Διεπουργική το Δεκέμβριο. Έτσι λοιπόν υπέθετα εφόσον αυτό το Κοινοβούλιο και αυτή η Επιτροπή την, από την περασμένη θητεία έχουν ζητήσει κάποιες αλλαγές στον κανονισμό λειτουργίας τον ίδιο του ΠΟΕ και δεν έχει γίνει τίποτα εν αναμονή της Ντόχα. Και εφόσον την Ολομέλεια της προάλλες, ουσιαστικά ψηφίσαμε κι εμείς και βάλαμε την ταφόπλακα πάνω στην Ντόχα, λέγοντας ότι τίποτα δεν προχωράει. Εάν δεν υπάρχει καμία αλλαγή στον ΠΟΕ, θα πρέπει μάλλον αυτή η Επιτροπή να αναθέσει στον Πρόεδρό τη να συντάξει μια επιστολή, να καλεί την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζητήσουν και από τους υπόλοιπους partner, τους εταίρους των διεθνών εμπορικών σχέσεων, να καθίσουν σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων και να αλλάξουν επιτέλους τον τρόπο λειτουργίας του ΠΟΕ. Χωρίς ε, να σημαίνει ότι θα, το κείμενο που έχουμε συντάξει θα είναι μια ωραία δήλωση προθέσεων, αλλά δεν θα αλλάξει την πραγματικότητα την οικονομική που γίνεται όλο και τραγικότερη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Χάμος από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Στέρντι ο οποίος ε, θέτει κάποια στοιχεία που βοηθούν πολύ τη συζήτηση. Πιστεύω και εγώ ότι έτσι μπαίνουμε σε μια ζωτική σημασία συζήτηση που έχει να κάνει με τις αρχές του διεθνούς εμπορίου και με τις ε, εξελίξεις του εν μέσω οικονομικής κρίσης. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πραγματικά και εδώ συμφωνώ με τον κύριο Στέρντι, χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε αυτό το καυτό θέμα. Γιατί τι είναι μη δεσμολογικό φραγμός και τι είναι. Τι είναι και τι δεν είναι. Και δεδομένου ότι δεν έχουμε σαφή εξήγηση από τον ΠΟΕ, κανείς μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικές προσεγγίσεις. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε το χρόνο μας, να μην βιαστούμε, ώστε ως Επιτροπή να λύσουμε τέτοια θέματα. Έχοντας κοιτάξει λίγο το πρώτο σχέδιο, κύριε Στάρντι, που μας προτείνεται, βλέπω κάποιες ανισορροπίες στην αιτιολογική σκέψη, στην αιτιολογική έκθεση, συγγνώμη, όπου περιγράφεται την διαφοροποίηση όταν προσπαθούμε να δώσουμε τον ορισμό των μη δασμολογικών φραγμών. Όμως τελικά δεν τη βλέπω αυτήν την διαφοροποίηση. Αν δείτε τα οικολογικά κριτήρια τα οποία έχουμε συζητήσει και εδώ στην Επιτροπή μας, όταν εξετάσαμε την έκθεση Ζαντό, ή... τα συζητήσαμε και με την έκθεση της κλπ, πολύ συχνά καταλήξαμε στη θέση ότι η επενδυτική μας πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη τέτοιους ε, παράγοντες που είναι μη δεσμολογικοί φραγμοί, οι οποίοι όμως αιτιολογούνται και αποτελούν και προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη. Έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα αποτελούν και μια διέξοδο για τις διάφορες ευρωπαϊκές οικονομίες ή γενικότερα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Στην Επιτροπή την Οικονομική ακριβώς συζητήσαμε πώς να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της ε, οικονομικής διακυβέρνησης και καταλήξαμε στο ότι πρέπει γενικότερα να βλέπουμε την οικονομική μας πολιτική και τις λύσεις που προτείνουμε. Λεβάνοντας υπόψη και άλλα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Γι' αυτό πιστεύω ότι χρειαζόμαστε χρόνο για να ξαναδούμε ολόκληρη την έκθεση και να δούμε τελικά πού ακριβώς πρέπει να επικεντρωθεί η Επιτροπή μας όσον αφορά αυτό το θέμα. Δύο παραδείγματα. Αν ε, δούμε το θέμα των περιβαλλοντικών αποφάσεων ε, που παίρνει η Ιαπωνία και που το συζητήσαμε στη, στα πλαίσια της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών με την Ιαπωνία. Κατά τη γνώμη μου, δεν πρόκειται πραγματικά για φραγμούς, έτσι όπως ε, το καταλαβαίνω, που πρέπει να ξεπεράσουμε. Όχι, πρέπει τις δικές μας επιδόσεις να βελτιώσουμε ως Ευρώπη για να ανταποκριθούμε ας πούμε μείωση διοξιδίου του άνθρακα κτλ. για να ανταποκριθούμε στα δικά τους τα κριτήρια έτσι όπως η απορνική αγορά τα αντιλαμβάνεται. Δεύτερον, και το έδωσε και κάποιος εδώ το παράδειγμα αυτό, η οδηγία REACH το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολύ συγκεκριμένη άποψη ότι πρέπει να εμείνουμε στο REACH και ότι το REACH δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως φραγμός. Άλλες χώρες όμως το βλέπουν σαν φραγμό. Θέλω να πω με αυτό ότι αυτά αποτελούν παραδείγματα σχετικά με τα οποία πρέπει να πείσουμε τους εταίρους μας να τα αντιμετωπίσουν ε, με πιο ανοιχτό πνεύμα, αλλά και εμείς να λάβουμε υπόψη μας τι ισχύει για τις δικές τους οικονομίες και γενικότερα για την οικονομία. Και πώς συνεισφέρουν τέτοια θέματα στο εμπόριο. Τέλος, θέλω να μας υπενθυμίσω, να υπενθυμίσω σε όλους μας το Aid for Trade. Και εδώ Υπάρχουν όμως κάποια εμπόδια. Οι οικονομικές επιδόσεις δεν ε, μπορούν να φτάνουν για πρόσβαση στην ε, Ευρώπη και στην ΕΚΟΝ το είπαμε ότι το εμπόριό μας πρέπει να συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη άλλων περιφερειών ή χωρών εταίρων μας. Άρα η επενδυτική μας πολιτική δεν αποτελεί μόνο ένα κομματάκι της εμπορικής μας στρατηγικής, δεν είναι κάτι εντελώς θεωρητικό, πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε, την επενδυτική μας πολιτική, μέσα σε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκτενέστερα το θέμα αυτό όσο συνεχίζονται οι διαδικασίες ομάδα μας θα υποβάλει σίγουρα κάποιες τροπολογίες στην έκθεσή σας. Ευχαριστώ κύριε Στέπη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόεδρος, ωραία, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Έχουμε εδώ τον κύριο Ντέρκοπο και ο Ποιος θα μιλήσει? Εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Ντούρκοπ. Mm. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει και την Επιτροπή σας και τον εισηγητή σας, όλους ιδιαίτερος, που ασχολείται με αυτό το θέμα των μη δασμολογικών φραγμών. Κάτι το οποίο δείχνει πόσο αποφασισμένοι είμαστε να αντιμετωπίσουμε τους μη δασμολογικούς φραγμούς και υπογραμμίζουμε τους διάφορους φραγμούς που εντοπίζονται μέσω εξέταση των διμερών αλλά και γενικότερων εμπορικών μας συμφωνιών. Ε, σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που εξετάζετε το θέμα αυτό και που θίγετε το εξής. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι με την απάλληψη των δασμών δεν εξακολουθούμε να υπονομεύουμε με μη ε, δασμολογικούς φραγμούς το εμπόριό μας. Από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μα αρέσει η περιγραφή των ε, διαφόρων περιπτώσεων που αναφέρονται στην έκθεση που δεν αντικατοπτρίζουν μόνο αυτά τα οποία λέμε εμείς στην έκθεσή μας, αλλά προσθέτουν και μια επιπλέον πτυχή. Θέλω όμως να υπογραμμίσω εδώ δύο πράγματα στις συστάσεις, που πιστεύω ότι είναι σημαντικά. Το ένα είναι το θέμα των προληπτικών ε, μέτρων. Όπως πολύ σωστά υπογραμμίζεται στην έκθεση, είναι ζωτική σημασία. Η εμπειρία μας διδάσκει ότι άπαξ και λαμβάνονται μέτρα μέσω νομοθετικής δράσης πολύ συχνά, είναι πολύ δύσκολο μετά να απαλλαγούμε από αυτά τα μέτρα. Άρα προληπτικά πρέπει να είμαστε σε θέση να αποφύγουμε τέτοιους φραγμούς να ισχύσουν. Έχουμε κάνει αρκετά, συνεργαζόμαστε στενά με τις αντιπροσωπείες μας που είναι οι κεραίες μας κατά κάποιο τρόπο, ο συνδετικός μας κρίκος με τους εταίρους μας για να δούμε τι ε, μέτρα σκοπεύουν να υιοθετήσουν οι εταίροι μας και από εκεί και πέρα ε, προσπαθούμε να πιέσουμε προς την κατεύθυνση που θέλουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ μπορεί να παίξει σίγουρα ένα πολύ χρήσιμο ρόλο, δεδομένου ότι εσείς συνομιλείτε με τους ομολόγους σας στις διάφορες αντιπροσωπείες που έχετε, οπότε λίγο πολύ αντιλαμβάνεστε τι, ρυθμίσει τι ρυθμίσεις σκοπεύουν να θετήσουν οι χώρες αυτές. Έπειτα, η συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να έχουμε feedback από τις επιχειρήσεις και να ακούμε και από αυτούς τι φραγμούς ε, μυρίζονται ότι θα αρχίσουν να ισχύουν. Γιατί βλέπετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί αλλιώς να έχει δίκτυο επαφών. Οι επιχειρήσεις έχουν αυτό το δίκτυο και είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν και οι επιχειρήσεις στις ε, εργασίες μας για να προβλέπουμε τα πιο σημαντικά εμπόδια που θα ισχύσουν. Κάτι άλλο για τις συστάσεις. Η σημασία των διεθνών προτύπων. Είναι πολύ σημαντικό, όπως έχουμε πει, ότι, στην ανακοίνωσή μας, ότι πρέπει να μπορούμε να αναπτύξουμε διεθνή πρότυπα. Να έχουμε κάποιο είδους εναρμόνιση, όπως τη λέμε, στη γλώσσα μας, ώστε οι κύριοι εμπορικοί μας εταίροι, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για νέους τομείς, ας πούμε ηλεκτρικά οχήματα, να μπορούν και εκείνοι να καταλαβαίνουν όπως και εμείς ποιοι πρέπει να είναι οι τεχνικοί κανόνες. Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Όχι, έχει να κάνει με ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό και πρέπει να συνεργαζόμαστε κι εμείς και με άλλα τμήματα και άλλε γενικές διευθύνσει τη Κομισιόν, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν τέτοιε διεθνεί προδιαγραφέ και πρότυπα. Κάτι τελευταίο τώρα για την σύσταση που έχει να κάνει με καλύτερη αξιολόγηση, καλύτερης ποιότητας αξιολόγησης. Έχετε διαπιστώσει ότι εμείς προσπαθούμε να έχουμε κάποια αξιολόγηση αντικτύπου για τις επιπτώσεις των ε, μη δασμολογικών φραγμών επί των επιχειρήσεών μας. Όμως καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κάποιος περιορισμός στο τι μπορούμε να κάνουμε. Δουλεύουμε με οικονομολόγους, με τον ΠΟΕ, με οικονομικά τμήματα, προσπαθώντας να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο, τον ποιοτικό αντίκτυπο των ε, μέτρων, των φραγμών. Ας πούμε, θα χαθούν θέσεις απασχόλησης. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνουμε αυτό, αλλά σημειώνουμε παρόλα αυτά τη σύσταση που κάνετε στην έκθεσή σας για να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως το μέτωπο αυτό. Για να συνοψίσω, η έκθεση κατά τη γνώμη μας δίνει μια νέα όθηση στην δικιά μας δουλειά για τους εμπορικούς φραγμούς. Είναι πολύ σημαντικό. Η επόμενη συζήτηση στο Συμβούλιο προβλέπεται αρχές Μαρτίου. Εννοείται ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο να έχουμε εγκεκριμένο το σχέδιο αυτό έκθεσης, οπότε οι συστάσεις θα μπορέσουν να συμπεριληφθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην επόμενη δική μα έκθεση. Να υπογραμμίσω επίσης ότι στις επόμενες εβδομάδε θα δημοσιεύσουμε τη νέα έκθεσή μας για τον προστατευτισμό, που επίσης έχει να κάνει με αυτό το θέμα των φραγμών. Έχουμε και την διάσκεψη του Νοεμβρίου, οπότε θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο το κείμενο αυτό προκειμένου να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας. Ο εισηγητής, ο Ρομπέρτ Αστέρντι, για τα τελικά του σχόλια. Ρόμπερτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θέλω εννοείται να περιορίσω ή να αναμειχθώ στα πρότυπα τα οποία μπορεί να υπάρχουν είτε από τον ΠΟΗ είτε οτιδήποτε άλλο στο οποίο αναφερθήκατε εσείς για τα ηλεκτρικά οχήματα για παράδειγμα, κάθε άλλο είναι προδιαγραφές που όλες οι χώρες παντού στον κόσμο πρέπει να τηρούν προς όφελος των καταναλωτών, του κοινού. Το στηρίζουμε απόλυτα λοιπόν. Κρίστοφερ, Εντάξει, καταλαβαίνω. Εκείνο πάει λίγο πιο μακριά από ό,τι εγώ, αλλά Κρίστοφερ, κοίτα. Η αρχική έκθεση έγινε ώστε να μπορούν διαφορετικοί άνθρωποι να πούν τις απόψεις τους. Καταλαβαίνεις ότι αν τα βάζαμε όλα μέσα χρειαζόμασταν τρεις τόμους. Όχι μια τέτοια έκθεση. Ήρθαν διάφοροι και μας είπαν τα προβλήματά τους και σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ξέρει τα περισσότερα από αυτά. Φυσικά και είναι καλή ιδέα να μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Αν έχουμε ένα τέτοιο σύστημα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν μη τι άλλο μπορούμε να το λέμε στην Επιτροπή. Κριστίν. Α, όχι. Ποιος ήταν, άλλος ήταν ο πρώτος. Ο Καντιέ. Έχει δίκιο. σε όλα. Όσον αφορά τους μη δασμολογικούς φραγμούς και άλλα. Μα εντάξει, υπάρχουν για ένα λόγο. Και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, το είπε και εκείνο, επιμένει για αυτούς. Φυσικά και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις προδιαγραφές μας, περιβαλλοντικές κλπ. Και να πείσουμε και άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά και θέλουμε να διατηρήσουμε τέτοιους φραγμούς για προφανείς λόγους. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τεράστια έκθεση για το ΡΙΤΣ, που βάζει προδιαγραφές για τις χημικές ουσίες και τα αγροχημικά. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για όλους εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν αποτελούν φραγμό για το εμπόριο. Είναι προκειμένου οι προδιαγραφές των άλλων να έρθουν στο ίδιο επίπεδο που είναι και οι δικές μας. Δεν ξέρω ποιος το είπε ο Κριστίν, έχεις δίκιο και συμφωνώ με όλα όσα είπες. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι και η Κριστίν και εγώ, μαζί με τον Πασκάλ Λαμί στον ΠΟΕ, στην ε, Υπουργική Διάσκεψη, το θέσαμε αυτό. Και εξετάζουμε τους κανόνες του ΠΟΕ για να δούμε τι αλλαγή πρέπει να γίνει σε αυτούς. Έχεις απόλυτα δίκιο πάντως, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Νομίζω ότι κάλυψα τα σημεία σας. Κοιτάξτε τώρα, δεν αντιτίθομαι στην ε, ιδέα ε, αυτή της ε, προστασίας, όχι μόνο των βιομηχανιών. Εγώ δεν είπα ότι είμαι εντελώ κατά τέτοιων μη δεσμολογικών φραγμών, εξαρτάται πώ χρησιμοποιούνται. Πρέπει να χρησιμοποιούνται για το σωστό λόγο και όχι να αποτελούν εμπορικό φραγμό. Έχουμε την κλασική περίπτωση της υποδηματοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπέφερε. Αν κάποιος παράγει υποδήματα ε, σε κόστος κάτω του κόστους του δέρματος, εντάξει προφανώς και πρέπει να υπάρχει κάποιος φραγμός στις αγωγές. Δεν είναι για να εμποδίσεις το εμπόριο είναι για να υπάρχει μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Είναι κάτι διαφορετικό. Αυτές τις αρχές πρέπει να τις έχουμε. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει ποτέ να υπάρχουν, γιατί μερικές φορές, όταν είναι για τη δημόσια υγεία, για παράδειγμα, για κάτι άλλο τέτοιο, να που Τώρα θέλω να επανέλθω λίγο σε αυτό που ακούστηκε πριν για το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Ναι, όλοι θέλα, θέλαμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να εξετάσουμε όπως θέλουμε την ε, έκθεση. Αλλά πρέπει να βιαστούμε για να επηρεάσουμε τα πράγματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι έτοιμο αν θέλουμε να μας ακούσουν. Γιατί κατά το παρελθόν δεν μας άκουγε η Επιτροπή. Τώρα, αν μη τι άλλο, δηλώνουμε τη θέση μας και εφόσον είμαστε έτοιμοι έγκαιρα μπορεί να μας ακούσει η Επιτροπή. Θα ακούσετε τις προθεσμίες σε λίγο και φροντίστε να υποβάλλετε τις τροπολογίες σας έγκαιρα γιατί θα θέλαμε να περάσει στην ε, Ολομέλεια του Δεκεμβρίου η έκθεση αυτή στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι 23, 23η αύριο δηλαδή στις 18, ε, 6 το απόγευμα. Και στις 11 ε, Οκτωβρίου ε, θα περάσει από την Επιτροπή. Σημείο 10. Πρόκειται για μία γνωμοδότηση για την ΑΦΕΤ που είναι η αρμόδια επιτροπή συστάσεις προς το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Εξωτερική ε, Υπηρεσία για τις διαπραγματεύσεις, εξωτερικής δράσης για τις διαπραγματεύσεις της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας. Θα πάει στην άφετο ο εισηγητής μας είναι ο Πάβελ Ζαλεύσκη που βρίσκεται εδώ και του δίνω και το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα πολωνικά. Πρόκειται για τη δεύτερη συζήτηση που κάνουμε για την ε, βρία αυτή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών με την Ουκρανία και ξέρουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η συμφωνία μια ιδιαίτερη συμφωνία. Ο στόχος εδώ δεν είναι μόνο το άνοιγμα της αγοράς, της Ουκρανικής αγοράς για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντίστροφα θέλουμε την οικονομία στην Ουκρανία να την αναδομήσουμε. Θέλουμε να ισχύουν στην Ουκρανία τα ίδια πρότυπα, διαδικασίες. Πρόκειται δηλαδή για τον εξυγχρονισμό της Ουκρανίας. Πρόκειται για μια συμφωνία όπου ε, περιλαμβάνει ένα μέρος της συμφωνίας σύνδεσης και σε αυτή τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών υπάρχουν κάποια τμήματα που όπως είπα ε, έχουν άμεση σχέση με τη Συμφωνία Σύνδεσης. Στις 19 Σεπτεμβρίου αποφασίστηκε ε, ε, άρχισε η νέα φάση των ε, διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με την Ουκρανία. Και εδώ θα ήθελα να ρωτήσω εδώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάτι. Πώς εξελίσσονται αυτές οι διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία για τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. Ακούσαμε κάποια θετικά πράγματα. Μας είπαν όμως ότι υπάρχουν και κάποια ίσονα προβλήματα τεχνικής φύσεως. Γι' αυτό και ρωτώ, τι περιμένει η Κομισιόν μετά από μια εβδομάδα διαπραγματεύσεων και τι προβλήματα παραμένουν ανοιχτά. Επίσης είναι πολύ σημαντικό κατά τη συζήτηση αυτή για τη Συμφωνία Σύνδεσης με την Ουκρανία όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ουκρανική Κυβέρνηση να συμμετέχουν ούτε μόνο τα κοινοβούλια, το Εθνικό του Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό. Και ο Ουκρανικός λαός πρέπει να συμμετέχει. Πήγα στην Ουκρανία και συνήντησα διάφορους εκπροσώπους της επιχειρηματικής ε, κοινότητας ε, της χώρας, με κυβερνητι... μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά και με ανεξάρτητους ειδικού που ενδιαφέρονται ε, για την ενσωμάτωση στην Ευρώπη της Ουκρανίας. Θέλω να σας ανακοινώσω κάποια σχόλιά τους, κάποιες προτάσεις τους, τις οποίες ενδεχομένως θα συμπεριλάβω την γνωμοδότηση ε, μέσα από τροπολογίες. Η προθεσμία λίγη αύριο. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η Συμφωνία Σύνδεσης θα πρέπει να λύσει παράλληλα ε, διάφορα προβλήματα στην Ουκρανία. Επίσης, πρόκειται για την επιστροφή του ΦΠΑ κατά την εξαγωγή των προϊόντων, τα οποία έχουν κατασκευαστεί στην Ουκρανία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Η κυβέρνηση της Ουκρανίας πολλές φορές προσπάθησε να λύσει το πρόβλημα, αλλά χωρίς επιτυχία μέχρι τώρα. Δεύτερον, οι τελωνιακές ε, διαδικασίες Τώρα, συνήθως, ε, η δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων που εισάγονται στην Ουκρανία, όλη αυτή η αξία ε, θα, είναι, θα ορίζεται πολύ ψηλότερη. Αυτό είναι κακό για τις ε, εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτον, προστασία των επενδύσεων και προστασία της ιδιοκτησίας στην Ουκρανία χρειάζεται. Ε, εξίσου πρέπει να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Τώρα, περνάω στις συναντήσεις μου με τους εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων και ανεξάρτητων ε, ειδικών επαγγελματιών και επιχειρηματιών και επαγγελματικών ενώσεων. Όλοι μου είπαν ξεκάθαρα ένα πράγμα κυρίως που θέλω να το τονίσω ιδιαίτερα εδώ. Υπάρχει η δυνατότητα, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, πριν από την επικύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης, βάση του άρθρου 217 παράγραφος 5, μπορεί λοιπόν το Συμβούλιο μετά από αίτημα της Κομισιόν να λάβει μία απόφαση που θα προβλέπει ότι μπορεί να αρχίσει να εφαρμόζεται η συμφωνία σύνδεσης πριν από τη θέση σε ισχύ του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί, διότι όλα δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών και τη Συμφωνία Σύνδεσης ε, θα ολοκληρωθούν πολύ γρήγορα. Ελπίζω ότι στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου να υπογραφούν οι συμφωνίες αυτές. Στο Κίεβο θα γίνει σύνοδος κορυφής το Δεκέμβριο και είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει την πρόταση αυτή. Εμείς ως Κοινοβούλιο θα στηρίξουμε την Κομισιόν, ώστε δηλαδή η Συμφωνία Σύνδεσης να αρχίσει να εφαρμόζεται άτυπα πριν από την επίσημη έγκριση του, αυτό, τη θέση σε ισχύ του. Αυτό είναι σημαντικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί η Συμφωνία Σύνδεσης είναι πολύ ευνοϊκή για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την Ουκρανία. Είναι πολύ σωστό δηλαδή η Ουκρανία να αρχίσει να λειτουργεί και να εφαρμόζει τις διατάξεις της Συμφωνίας Σύνδεσης εφόσον θα έχει υπογραφεί η Συμφωνία. Επίσης, τι άλλο έχω να σας πω, οικονομικά προβλήματα στην Ουκρανία. Επίσης, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας. Ε, όταν διαπραγματευόμαστε συμφωνία ελευθερών συναλλαγών με την Ουκρανία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η Ουκρανία μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να κάνει ε, μια μεταρρύθμιση του, της σημαντικότερης εταιρείας ε, αερίου της. Τώρα, τι εσκίαζε μέχρι τώρα τις διαπραγματεύσεις. Ε, ε, υπήρχε η πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία, η σύλληψη της κυρίας Γιούλια Τιμοσέγκο και υπάρχουν και κάποια εξωτερικά θέματα, δηλαδή η Ρωσία η οποία προσπάθησε να απομακρύνει την ε, Ουκρανία από την Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών και της πρόσφερε μια τελωνιακή ένωση η οποία θα περιελάμβανε και το Καζαχστάν και τη Λευκορωσία εκτός από Ρωσία και Ουκρανία. Εγώ έχω λάβει επίσημη άποψη εδώ, την άποψη του επιχειρηματικού κόσμου της Ουκρανίας, ε, μια πολύ σοβαρή επαγγελματική και επιχειρηματική ένωση της Ουκρανίας μου έστειλαν την επίσημη άποψή τους, όπως επίσης και κάποιοι ειδικοί που ενδιαφέρονται για την ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι αυτοί έστειλαν τις απόψεις τους που είναι ξεκάθαρες. Τα μέλη της κοινότητας των πολιτών θεωρούν ότι η Συμφωνία Σύνδεσης δεν είναι μόνο μια συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όχι. Είναι μια συμφωνία η οποία πραγματικά επηρεάζει βαθιά τη ζωή των Ουκρανών. Και με πολύ θετικό τρόπο μάλιστα, θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις, το εμπόριο, θα βελτιώσει δηλαδή τις εξελίξεις στους τομείς αυτούς. Και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών με τους οποίους συνομίλησα θεωρούν ότι η συμφωνία αυτή δεν πρέπει να πολιτικοποιηθεί αλλά να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό. Από την άλλη πλευρά μια ταχεία εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών θα θέσει σε σωστές βάσεις τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας. Αναφέρομαι εδώ κυρίως στις οικονομικές σχέσεις. Θα επηρεάσει τις οικονομικές σχέσεις βέβαια και θα τις βάλει σε σωστή βάση τις οικονομικές σχέσεις, τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Αυτά ήθελα να πω και περιμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Κάθε θέμα είναι πολύ σημαντικό και αυτό επίσης, αλλά ε, πρέπει και να προχωρήσουμε. Ο επόμενος ομιλητής μας είναι ο Τζόρτζ Κούτας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας θα εδρεώσει τις πολιτικές σχέσεις και την οικονομική ενσωμάτωση μεταξύ των δύο εταίρων, την οικονομική ολοκλήρωση. Η Ουκρανία προσχώρησε στον ΠΟΕ το 2008 και αυτό διευκόλυνε τις συζητήσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας. η Ουκρανία θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία για το εμπόριο. Εδώ μιλάμε για οικονομική συνεργασία, ενεργειακή, ε, συνεργασία στην ασφάλεια, στον τομέα των θεωρήσεων κλπ. Όλα αυτά τα έχει αναφέρει ο κύριος Ζαλεύσκη και γι' αυτό τον συγχαίρω για το έργο του. Πιστεύω ότι πρέπει να προσέξουμε περισσότερο όταν μιλάμε για την ενεργειακή ασφάλεια. Είναι ε, χώρα μετάβασης ε, η Ουκρανία, γιατί από εκεί περνάει το ρωσικό φυσικό αέριο και όλοι ξέρουμε ότι το 2009 η κρίση στο φυσικό αέριο επηρέασε τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Δυστυχώς οι ευρωπαϊκές πολιτικές ε, τώρα βρίσκονται εκτός τομέα ενέργειας γιατί κυρίως ε, ε, προωθούν πολιτικούς στόχους. Και έτσι δεν έχουμε πρόσβαση σε εξωτερικές πηγές φυσικού αερίου. Εδώ όμως ε, μπορεί να αποβεί πολύ καλό εταίρος η Ουκρανία. Πιστεύω ότι πρέπει να λύσουμε λοιπόν τα προβλήματα με την Ουκρανική νομοθεσία. Δεν υπάρχουν αρκετοί νόμοι που ρυθμίζουν τους τομείς πετρελαίου και αερίου. Γι' αυτό λοιπόν η απόκτηση αδειών, για παράδειγμα, ε, ε, η αδειοδότηση πρέπει να είναι διαφανή διαδικασία. Πιστεύω ότι η Ουκρανία έκανε σημαντικά βήματα για να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό επιβεβαιώνεται από τη δήλωση του Πρωθυπουργού της Ουκρανίας τον Αύγουστο. Είναι υπέρ της προοπτικής της ε, συμφωνίας σύνδεσης σε βάρος της Τελωνιακής Ένωσης που πρότεινε η Ρωσία Πιστεύω ότι χρειάζεται κάποια πρόοδο σε ορισμένους τομείς όπως προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών ελευθεριών, ε, πρότυπα εργασίας, προαγωγή αξιοπρεπούς εργασίας, κατάργηση διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών. Θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες και δυστυχώς ο χρόνος πιέζει πολύ. Ελπίζω να είναι μια καλή γνωμοδότηση μετά από τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ. Έχω αρκετούς που ζητούν το λόγο για να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. Θα έχουμε περιορισμό χρόνου από εδώ και πέρα. Τρία λεπτά με το ρολόι. Ο Ντάνιελ Κάσπαρη, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή. Δεν είναι αυτονόητο ένας εισηγητής από την Επιτροπή αυτή να βρει χρόνο τακτικά να ε, συνομιλεί με τους εταίρους ε, από διάφορες χώρες. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε ευγνώμονες επίσης διότι και στο σχέδιο γνωμοδότησης και στην παρουσίαση σήμερα κατέστη σαφές ότι εδώ πρόκειται κυρίως για το εμπόριο, γιατί έχω την εντύπωση ότι τις τελευταίες εβδομάδες υπήρχε η απειλή ε, πίσω από το σημαντικό θέμα δημοκρατία κράτους δικαίου κλπ. Ε, να υποβαθμιστεί το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας. Και είμαι ευγνώμων στον κύριο Ζαλεύσκη ο οποίος ανέδειξε τα οικονομικά προβλήματα και τις προκλήσεις στον τομέα αυτό. Ιδιαίτερα τη διπλή, διπλές τιμές, διπλή τιμολόγηση, ε, επιστροφές και, και λοιπά. Αυτά θα πρέπει ε, να πούμε ότι σε σημαντικό βαθμό έχουν λυθεί, αλλά πολλά μέλουν ακόμα να γίνουν. Επίσης ε, η υπόθεση Τιμοσέγκο βαραίνει πολύ την, ε, τις σχέσεις με τις χώρες αυτές, σίγουρα, αλλά μην πούμε κιόλα ότι θα περάσει η συμφωνία αυτομάτως σχεδόν μόλι λυθεί η υπόθεση Τιμοσέγκο. Όχι. Θα πρέπει να τα δούμε αυτά, πρέπει να εντατικοποιήσουμε τι οικονομικέ σχέσει. Αυτό είναι το αντικείμενο τη συμφωνία. και εκεί θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά και το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ω προ τι οικονομικέ παραμέτρου τη συμφωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για την ε, συντομία, ο Χέλμουντ Σόλτς από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη και ευχαριστώ τον εισηγητή για το κείμενό του αλλά και για τις παρατηρήσεις που έκανε σήμερα για το σημαντικό θέμα αυτό ε, της εμπορικής διάστασης αυτής της συμφωνίας σύνδεσης που είναι και κομμάτι της ε, Πολιτική γείτονα προ του ανατολικούς γείτονε, θεωρώ εγώ. Είναι σημαντικό. Γιατί αυτό θα προδικάσει και τη συμφωνία στο μέλλον με την Ουκρανία. Δύο πράγματα θέλω να τονίσω ιδιαίτερα που πρέπει να αναδειχθούν περισσότερο στη νομοδότηση. Πρώτον, η σχεδιαζόμενη ε, ζώνη, η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Συμφωνίας Σύνδεσης για να μην γίνουν κινήσεις αποσύνδεσης των δύο αυτών συμφωνιών. Αυτό από την αρχή πρέπει να το ε, αποκλείσουμε. Πρέπει λοιπόν να, θεωρεί, να θεωρείται μια ενιαία προσέγγιση αυτή. Αν το 80% των νομοθετικών διατάξεων σε όλους τους τομείς ε, ε, είναι τώρα αντικείμενο διαπραγματεύσεων στα πλαίσια του κοινοτικού εκτιμένου, καταλαβαίνετε πόσο τεράστια είναι η πρόκληση για τη χώρα αυτή. Θα ήθελα λοιπόν και εμείς ως Επιτροπή να τονίσουμε ότι αναλαμβάνουμε μία ευθύνη και για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ε, ανάπτυξη και τη σταθερότητα στην Ουκρανία. Είχαμε πει την τελευταία φορά ότι βεβαίως η Ουκρανία ε, βρίσκεται σε μια σύνθετη κατάσταση και θα είναι και στο μέλλον όταν θα πάει να εφαρμόσει όλες αυτές τις νομικές διατάξεις. Και εμείς μέσα από την οικονομική συνεργασία θα πρέπει να δώσουμε τη συμβολή μας ώστε να μην αποσταθεροποιηθεί η πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία. Τώρα, δεν ξέρω αν τα χρονοδιαγράμματα είναι ρεαλιστικά. Είπαμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θέλουμε πριν από τη θέση σε ισχύ κάποιων συμφωνιών να αποφανθούμε και θα πρέπει να ε, ενημερωθούμε για τα αποτέλεσματα των διαπραγματεύσεων και να ακούσουμε και τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Αυτά λοιπόν θα κοιτάξουμε να αναδείξουμε μέσα από τροπολογίες και κατά τα άλλα πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία με τον εισηγήτη. Ευχαριστούμε. Από το ΕΛΚΟ κυρίως ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Γκλάτφελντερ. Για, για τα εμπορικά ζητήματα, ιδίως για τις εμπορικές πτυχές των γεωργικών προϊόντων. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το πλαίσιο, διότι η Ουκρανία έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες ε, παραγωγής. Και επειδή υπάρχουν ε, και κοινά σύνορα, οι εμπορικές σχέσεις κάποιες φορές αντί να διευκολύνονται παρεμποδίζονται. Οπότε Υπάρχουν και τέτοιου είδου επιπτώσει. Σε ό,τι φορά λοιπόν τα αρχικά ζητήματα, η Ουκρανία είχε αναφέρει το θέμα των εγγύσεων. σίγουρα. Υπάρχουν ε, περισσότερο ευαίσθητα προϊόντα, ιδίω τα δημετριακά. και ιδίω εάν εξαιτία αυτού του τομέα υπήρξε, υπήρξε, υπήρχε αύξηση των εκπομπών στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα καταλήγαμε σε έλλειψη ισορροπία λοιπόν και δύσκολα θα καλυπτόνταν οι ανάγκε τη Ευρωπαϊκή Αγορά, Σε ό,τι αφορά τη ζάχαρη, Πρέπει να διευκολυνθούν εισαγωγέ, γιατί είμαστε σοβαροί εισαγωγή, άμεση εισαγωγή ζάχαρη. Η συνέπεια λοιπόν θα μπορούσε να είναι ε, ότι κάποια προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες περνώντας από την Ουκρανία τελικά να μην ανταποκρίνονται στις δικές μας τις προδιαγραφές και να καταλήγουν στην ευρωπαϊκή αγορά παρόλα αυτά. Αυτό θα πλήξει τη σταθερότητα της διεθνούς αγοράς ζάχαρης. Τέλος, σε ό,τι αφορά την ευζοία των ζώων, στην Ευρώπη έχουν γίνει τεράστιες επενδύσεις γι' αυτό. Όπως την ευζοία των ε, οτοκών ορνηθών στην Ουκρανία. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους μέτρα. Οπότε προϊόντα που προέρχονται από αυγά ή και τα ίδια τα αυγά μπορεί να εισάγονται στην Ευρώπη με χαμηλότερο επίπεδο και αυτό πλήττοντας τους Ευρωπαίους παραγωγούς που έχουν αναλάβει και το πρόσθετο κόστος για να εξασφαλίσουν ακριβώς την κάλυψη των μέτρων ευζοίας των ζώων. Επιπλέον ενώ στην Ευρώπη υπάρχουν τέτοιου είδους μέτρα και καθώ στι τρίτε χώρε δεν υπάρχουν, θα έπρεπε τα προϊόντα αυτά να τα αντιμετωπίζουμε ω ευαίσθητα, ιδιαίτερη κατηγορία. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Κυρία Κοχμερίν, από την Άλντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλώ να ευχαριστήσω την, τον εισηγητή για την προσέγγιση του. Δεν έχω πολλά να προσθέσω σε όσα είπατε και επισημάνατε, διότι Κάνατε μια πολύ καλή μελέτη του θέματος. Απλώς σίγουρα η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου και Σύνδεση είναι πολύ σημαντική, διότι η Ουκρανία και ως εταίρος και ως γειτονές αποτελεί ήδη από μόνη της μια πρόκληση. Είναι μια χώρα την οποία θέλουμε να την τραβήξουμε πιο κοντά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα υπάρχουν και οικονομικά ωφέλη που μπορεί κανείς να αντλήσει από αυτή τη σχέση. Και για τις δύο πλευρές. Θέλουμε λοιπόν η Επιτροπή να μας πει αν έχει επιτελεστεί πρόοδο για εκκρεμή ζητήματα. Ζητήματα που ήταν αφιλεγόμενο τώρα. Επίσης, αναφέρθηκε ότι χρειάζεται αναδιάρθρωση και εξυγχρονισμό της Ουκρανίας εν γέννη. Αυτό θα είναι δύσκολο από άποψη πολιτικής ισορροπία. Και η δική μα ομάδα ασχολείται με ζητήματα και εκδημοκρατισμού και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ή άλλως. Αυτά τα θεωρούμε λοιπόν ύψης της σημασίας. Αλλά και η σχέση με τη Ρωσία. Αυτό παραμένει μείζον ζήτημα. Θα ήθελα λοιπόν να δω κατά πόσον μπορούμε να τηρήσουμε εδώ την προθεσμία που προβλέπουμε. Το τέλος της φετινής χρονιάς. Εάν δούμε τους περασμένους χειμώνες, οι αναμνήσεις που μας έρχονται τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε τότε μας δείχνουν ότι το τέλος Σεπτεμβρίου θα είναι κρίσιμο ορόσημο. Χρειάζεται να επιτελεστεί επί... κατεπηγόντως πρόοδος τις ερχόμενες εβδομάδες. Και, Πρόεδρε, θα μιλήσω και γερμανικά γιατί απευθύνομαι και στον κύριο Κασπάρη. Ε, όπως είπα και στον ίδιο, η κατάσταση και η εξέλιξη των νομικών ε, διαστάσεων είναι ζητήματα που θα πρέπει να καλύπτει η έκθεση. Είναι σημαντικό λοιπόν και αυτό να το λάβουμε υπόψη, αλλά είμαι αισιόδοξη. Ο εισηγητή μα θα το πετύχει με τρόπο συνεπή. Και έτσι θα καταλήξουμε σε αίσια έκβαση. Ευχαριστούμε. Και τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι εξελίξεις υπάρχουν από τις διαπραγματεύσεις. Ο κύριος Λεπισόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω όσα υπόθηκαν από τους ε, συναδέλφους σας και τον κύριο Ζαλεύκη. Από την άποψη της Επιτροπής συμμεριζόμαστε απόλυτα τις απόψεις που εκφράστηκαν. Και τις παρατηρήσεις που έγιναν, απλώς μερικές συμπληρώσεις. Κύριε Ζαλεύκη, συμφωνώ μαζί σας, πέραν ενός σημείου. Δεν μπορούμε να υπογράψουμε τη συμφωνία ακόμη αν και από πολιτικής άποψη στόχο μας είναι ο Δεκέμβριο. και στο επίπεδο της Συμφωνίας Σύνδεσης. Συμφωνούμε λοιπόν απολύτω με όσα υπόθηκαν για το πώς αντιμετωπίζουμε την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών και τη Συμφωνία Σύνδεσης. Κάτι που τουλάχιστον δύο φορέ σχολιάστηκε για την ενέργεια. Γι' αυτό έχω να σα πω το εξή. Σύντομη ανασκόπηση τη χθεσινή συζήτηση. Χθες ο Επίτροπος Εμπορίου δήλωσε στον αντιπρόεδρο της χώρας ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία με την Ουκρανία εάν το κεφάλαιο της ενέργειας δεν εξασφαλίσει ότι θα αποφύγουμε τις κρίσεις του παρελθόντος, της τελευταίας διετίας ιδίως. Αυτό είναι κάτι στο οποίο είμαστε μετακίνητοι. Η Ουκρανική πλευρά το δέχεται. Οπότε θα μπορέσουμε να οδεύσουμε και προς μια συμφωνία σχετικά. Σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, τη γεωγρα... γεωστρατηγική διάσταση της συμφωνίας. Το έχουμε όλοι κατά νου. Το Ουκρανικό Κοινοβούλιο υιοθέτησε κείμενο που αναφέρεται στη σχέση συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή, στην ε, σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την καλή σχέση συνεργασίας με τη Ρωσία έπειτα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από του πολιτικού ηθήνοντε τη χώρα. Και επειδή περνάει γρήγορα η ώρα, σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει αυτέ καθε αυτέ, όπω είπα προηγουμένω, υπήρξε διευπουργική χθε μεταξύ του Επιτρόπου Γκεχβίρτ, Επιτρόπου Εμπορίου και του Επιτρόπου Γεωργία και του Αντιπροέδρου Κλούγεφ. Η διευπουργική αυτή συνάντηση είχε πολύ θετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερω επειδή η Ουκρανική πλευρά αποδέχτηκε τις δικές μας κόκκινες γραμμές. Σημεία στα οποία παραμένουμε αμετακίνητοι στις διαπραγματεύσεις, όπως ε, το θέμα της ενέργειας. Θα υπάρξει κεφάλαιο πλήρες για τα θέματα της ενέργειας, τα γεωργικά προϊόντα, αναφέρατε εσείς λόγου χάρη τη ζάχαρη. Εμείς πλαισιώσαμε τις παραχωρήσεις μας στο επίπεδο της ζάχαρης λόγου χάρη για να αποφύγουμε περιπτώσεις όπως αυτές που ανέφεραν οι βουλευτές, δηλαδή την ε, κυκλική κυκλοφορία της ζάχαρης και την εμπορία της μέσω της Ουκρανίας από τρίτες χώρες. Σε βιομηχανικό επίπεδο έχουμε σημαντική παραχώρηση από την Ουκρανική πλευρά για την απελευθέρωση της αυτοκινητοβιομηχανίας και με αυτό θα κλείσω, Πρόεδρε. Πολύ θετική συνάντηση χθε, η διευπουργική, και θα προλάβουμε, πιστεύω, να τηρήσουμε τι προθεσμίε που ανέφεραν όλοι σα οι συνάδελφοι στη συζήτηση. Θα έχουμε συμφωνία στο τέλο τη χρονιά, πιστεύω. Πρόεδρο. Ωραίε ειδήσει αυτές. Κύριε Ζαλεύσκη, τελικές παρατηρήσεις. Πρόεδρε, για να απαντήσω σε ορισμένα από τα σημεία που έθιξαν οι συνάδελφοι. Ο κύριος Κούτας μίλησε για τη σημασία της Ουκρανίας και το ρόλο της στον ΠΟΕ. Ήταν ένα πρώτο βήμα πολύ σημαντικό για την ε, απελευθέρωση του εμπορίου. Η προσχώρηση της Ουκρανίας επιτρέπει και ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά της χώρας αυτής. Η συμφωνία θα μας επιτρέπει να κάνουμε ακόμη πιο εύκολη την πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όσο για την διαφανή ε, λειτουργία του κρατικού συστήματος, του κρατικού μηχανισμού της Ουκρανίας, αυτό είναι καθοριστική σημασία. Σημειώνω σε είπε ο συνάδελφο Κασπαρία, καθώς και συνάδελφο Κοχμερίν, γιατί πέραν αυτού υπάρχει και το θέμα των ε, δικαιωμάτων των πολιτών, ο σεβασμός των δικαιωμάτων αυτών, που κάποιε περιπτώσεις παραβιάζονται, όπως στην περίπτωση Τιμοσέγκο, είναι θεμελιώδου ε, σημασία για τις δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης δεν είναι το πρόβλημα μόνο οι πολιτικές απαγορεύσεις αλλά και η ελεύθερη άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων λόγω χάρη. Είναι ένα θέμα που σε εμά ως βουλευτές είναι προσφυλέ προφανώς Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ακούμε και την Επιτροπή να λέει ότι θα πετύχουμε κάποιες ε, εγγύησεις για τη μεταφορά του ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ανατολική Ευρώπη και προς τις μας. Αυτό για μας έχει ιδιαίτερη αξία. Είναι κάτι που ευτυχώ το κατανοεί η Ουκρανική πλευρά. Όμως, οφείλουμε να πούμε ότι βρισκόμαστε στην δημιουργία ενός δεσμού ηθικού πέραν όλων των άλλων διαστάσεων με την Ουκρανία. Η συνεργασία μας με την Ουκρανία περνάει και από την επιρροή της Ρωσίας που αποθαρρύνεται να υπογράψει εμπορικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως ό,τι φορά το φυσικό αέριο. Εκεί θα μπορούσαν να υπάρξουν ε, και νέες διενέξεις στο μέλλον. Έτσι λοιπόν θα πρέπει με τρόπο πολύ ευθύ και αποφασιστικό να τηρήσουμε μια συγκεκριμένη στάση, ότι δηλαδή μπορούμε να ζητάμε πράγματα από την Ουκρανία, αλλά και να τη στηρίξουμε, εφόσον πολλές φορές η Ουκρανία αγοράζει φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Οι τιμέ είναι πολύ πιο ψηλέ για την Ουκρανία από ό,τι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε λοιπόν γιατί συμβαίνει αυτό. Όταν μιλούμε για δασμολογικά ζητήματα στις διαπραγματεύσει. Η Ουκρανία θα χρειαστεί λοιπόν τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να εξομαλυνθούν οι σχέσεις της με τη Ρωσία σε ό,τι αφορά την εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Ουκρανική επικράτεια. Άλλο σημείο. Το σχολείο ο συνάδελφο Σόλτ. Δυνατότητα υλοποίησης, πραγμάτωσης των στόχων. Όχι δηλαδή μόνο διαπραγμάτευση της συμφωνίας, αλλά και μεταφορά της συμφωνίας στην πράξη. Οι εμπειρίε μα ω τώρα δεν ήταν ε, οι πιο ρόδινε, διότι η Ουκρανία ω τώρα έχει προσυπογράψει αρκετέ συμφωνίε, έχει προσυπογράψει δηλώσει, αλλά μετά χρονοτριβεί ιδιαίτερα για την ε, πραγματοποίηση των στόχων στην πραγματικότητα. Έτσι από τώρα πρέπει να διερωτηθούμε. Σκοπεύει να δώσει ηλική υπόσταση στις συμφωνίες αυτές η Ουκρανία. Με τις σημερινές κρατικές δομές, ε, με τους φορείς και τις επιτροπές που υπάρχουν ε, και σε άλλες χώρες, στην Πολωνία, δεν μπορεί να διευκολυνθεί η Ουκρανία στο να μεταφέρει το ευρωπαϊκό κεκτημένο αλλά ακόμη και τα οικονομικά μέσα για την Ουκρανική πραγματικότητα σε σχέση με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να βελτιωθούν. Υπάρχουν λοιπόν ε, πολλά περιθώρια να θεσπιστούν ακόμη περισσότερα μέτρα για την επόμενη χρονιά. Να κλείσουν λοιπόν γρήγορα οι διαπραγματεύσει, αλλά να προβλέπονται και τα επόμενα βήματα. Η θέση σε ισχύ της συμφωνίας, ε, της προσωρινής συμφωνίας είναι σημαντική, να είναι άμεση, αλλά θέλουμε να επαγρυπνήσουμε και για την ε, πραγματική υλοποίηση της συμφωνίας. Όσο για τον γεωργικό τομέα, υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει μεγαλύτερη απελευθέρωση για τα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από την Ουκρανία και των υπολείπων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω μεταξύ των διαφορετικών αυτών ε, προτιμήσεων έχει πετύχει ένα καλό σημείο ισορροπίας. Διότι η Ουκρανία νομίζω ότι μεταξύ πολλών χωρών παγκοσμίω έχει από τι μεγαλύτερε δυνατότητε αύξηση των γεωργικής τη παραγωγή. Μιλάμε πολύ πλέον για την επισητιστική ασφάλεια. Ο ρόλο τη Ουκρανία εδώ είναι κέριο. Μεταξύ του CFTA τη συμφωνία δηλαδή ελεύθερου εμπορίου, μπορεί να πετύχει η σταθεροποίηση τη γεωργική τη παραγωγή η Ουκρανία, βελτίωση και μπορεί να παρέχει στην ε, παγκόσμια αγορά καλύτερα προϊόντα. Το θέμα Τιμοσέγκο. Ναι, ναι, ολοκληρώνω. Το ζήτημα αυτό πρέπει να επιληθεί με τρόπο φιλίσχο και ειρηνικό. Είναι γνωστή η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα βρεθεί λύση τις προσεχείς εβδομάδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Την έχετε την γνωμοδότηση. Προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών είναι αύριο στις 6 το απόγευμα. Πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα στα επόμενα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε την ανταλλαγή για το θέμα 13 που θα μας πάρει πιο πολύ χρόνο. Οπότε στα επόμενα να είσαστε σύντομοι. Σημείο 11 στην ημερήσια διάταξη. Είναι γνωμοδότηση για την ΑΦΕΤ. Συστάσεις στο Συμβούλιο και την Επιτροπή για τις Διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωργία για τη Συμφωνία Σύνδεσης. Ε, είναι κάτι παράλληλο με το θέμα της Ουκρανίας. Ε? Έχετε την, ε, το σχέδιο γνωμοδότησης στους φακέλους σας. Δεν είναι εδώ όμως ο σύγκητής. Κασπάρη ποιος. Όχι κύριε Κασπάρη δεν. Ποιος θα την αντικαταστήσει κάποιος άλλος. Ο κύριος Στάστνη. Ευχαριστώ. Η κυρία Αντρίκιενε δεν κατάφερε να είναι εδώ, όπως ξέρουμε. Ο κύριος Κάσπαρ όμως χρειάστηκε να φύγει, οπότε με άφησε εμένα να αναλάβω αυτό το θέμα και θα φροντίσω να είμαι και σύντομος, όπως είπατε. Η Γεωργία, όπως ξέρουμε, αποτελεί σημαντικό εταίρο στην περιοχή. Είναι μια χώρα η οποία έχει πετύχει τη μεγαλύτερη πρόοδο όσον αφορά τη δημοκρατία, την ανοιχτή κοινωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρουμε ότι για την Γεωργία αποτελεί τον πιο σημαντικό εμπορικό εταίρο. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό για αυτούς και είναι σημαντικό και για μας να συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Γεωργία έχουν ήδη συμφωνία συνεργασίας από τον Ιούλιο του 1999 και μετά έχουν και διμερή συμφωνία που μιλάει για μια εμπορική συμφωνία σε βάθος και ανοιχτή. Η συμφωνία αυτή είναι πολύ σημαντική για τη Γεωργία, η οποία θέλει να ενισχύσει τις εμπορικές της σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς, δεν έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος τελευταία. Όλες οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν ε, τον ε, Ιούλιο για το DCFTA. Όμως, όπως ξέρουμε, δεν υπάρχει πρόοδος όσον αφορά δηλαδή την εκτενή και ολοκληρωμένη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Ελπίζουμε να επιτευθεί κάποια πρόοδος και η κυρία Αντρίκιανε είναι στη διάθεσή μας προκειμένου να φανεί η σημασία που έχει αυτή τη εκτενούς και ολοκληρωμένη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία. Είναι πολύ σημαντικό και απέναντι στους ανατολικούς εταίρου μας. Η Γεωργία είναι μια χώρα παρά την σύγκρουση που έλαβε χώρα εκεί πρόσφατα. Ξέρουμε ότι οι πολίτες εκεί είναι από αυτούς που χαίρουν τις μεγαλύτερες ελευθερίες στο κράτος τους σε σχέση με αλλού. Αποτελεί λοιπόν μία από τις βασικές προτεραιότητες και της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, δύο λεπτά ο καθένας τώρα. Παρακαλώ, ο επόμενος. Ευχαριστώ πολύ. Όπως και με την Ουκρανία, έτσι και εδώ μπορούμε να πούμε ότι η Γεωργία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στρατηγικά μας ενδιαφέρει η περιοχή προκειμένου να διασφαλίσουμε εκεί σταθερότητα και ευημερία στη χώρα, λέει ο κύριος Κιούτας. Συνεπώς μια τέτοια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών θα ενισχύσει κάτι τέτοιο. Η Γεωργία είναι στο σωστό δρόμο. Παρ' αυτά επιδέχεται ακόμα βελτιώσεις. Εξού και οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξάλλου. Αναφέρομαι κυρίως στο θέμα των ε, τεχνικών φραγμών, το θέμα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ. Πιστεύω επίσης ότι η Γεωργία πρέπει να προσφέρει τους πόρους που χρειάζονται για να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις της στο νομοθετικό και το δικαστικό τομέα, προκειμένου να προσαρμοστεί στι απαιτήσει μια εκτενού και ολοκληρωμένη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών DCFTA. Πρέπει να φροντίσουμε επίσης να υπάρχει καλός έλεγχος των προδιαγραφών για τα προϊόντα της. Με τις δικές μου τροπολογίες θα προσπαθήσω να υπογραμμίσω τη σημασία που έχει το δίκαιο εμπόριο, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι συνθήκε εργασίας, η χρηστή διακυβέρνηση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για την Συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ για τη συμφωνία σύνδεση, δηλαδή. Ευχαριστώ. Κυρία Μουσκαρδίνη. Σύντομα, Πρόεδρε, πιστεύω ότι για όλες τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που επέβαλε στις χώρες αυτές ε, με το ζόρι κάποια πράγματα, θα πρέπει να τις πλησιάσουμε. Να αναπτύξουμε μαζί τους νέες σχέσεις, εμπορικές καταρχάς και να γίνει μια καινούργια αρχή, κοιτάζοντας σε πρώτη φάση το πρόβλημα των γεωργικών προϊόντων. Εφόσον είμαστε βέβαιοι, θα πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρξει περίπτωση επεξεργασίας ή περάσματος τοξικών προϊόντων, τοξικών μάλλον ουσιών, επειδή υπήρξαν πυρηνικές δοκιμές στο έδαφος της χώρας αυτής. Θα πρέπει έτσι να επιταχύνουμε την επίτευξη συμφωνίας για να μπορέσουν αυτές οι χώρες να βοηθηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταρτήσουν τις κατάλληλες πολιτικές σε μερικά χρόνια να μην βρεθούμε να αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα που κανείς δεν έθιξε. Ένα πρόβλημα που και για τις χώρες ε, στην επικράτεια των οποίων υπάρχουν τέτοια προβλήματα είναι επιζήμιο και για τους ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έχουν καταναλώσει αυτά τα προϊόντα εντωμεταξύ. Πρόεδρος. Και τώρα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Κουσόλ. Πιο γρήγορος από ό,τι για την Ουκρανία θα είμαι τώρα, Πρόεδρε. Συμφωνώ κατά πολύ με όσα είπαν οι συνάδελφοι βουλευτές. Απλώς κάποιες ε, παρατηρήσεις πιο συγκεκριμένες για όσα σχολιάστηκαν, αλλά θα τα πω δημερώς τους ενδιαφερόμενους. Για αυτή τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Γεωργία, να πω ότι όπως και για την Ουκρανία υπάρχει ατζέντα μεταρρυθμιστική που θα πρέπει να φέρει εις πέρας η χώρα αυτή και όταν θα έχει προχωρήσει αρκετά στις μεταρρυθμίσεις, τότε θα συζητήσει περισσότερο εντατικά μαζί μας για τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών, το είπε ο κ. Σόλτς προηγουμένως και για την Ουκρανία. Παρομοίως και εδώ αφορά το κοινοτικό και εκτιμένο εδώ η σχέση αυτή, διότι μιλάμε για οικονομική ολοκλήρωση. Σας καλώ να παρακολουθήσετε τη σύνοδο Eastern Partnership, εταιρική σχέση προς με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών ε, εκπροσώπων και των ανατολικών αυτών χωρών και εκεί θα ακούσουμε και τη Γεωργία. Θα δούμε κατά πόσο είναι πρόθυμη να πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις που τις έχουν ζητηθεί από εμάς. Τότε πολύ γρήγορα θα ολοκληρωθεί η εξέταση της συμφωνίας τους προσεχείς μήνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο εισηγητής για τελικές παρατηρήσεις. No Δεν υπάρχουν. Very quickly, as I... Πολύ γρήγορα. Ακούγοντα, ε, σημείωσα όλα τα σχόλια. Ευχαριστώ στου συναδέλφου, αλλά από τα έγγραφα γνωρίζω και η κυρία Αντρικένε, ξέρω ότι θα συμφωνούσε, ότι η Γεωργία έχει τις τεχνικές προϋποθέσεις για να μπορεί να συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών Και όπω είπε και η κυρία Μοσκαρντίνη, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, να δούμε τι πρόοδο επιτελείται. Αλλά τα τελευταία χρόνια υπήρξαν πολλέ έλεγχε στη Γεωργία, οπότε νομίζω δεν θα υπάρξουν δυσκολίε να διεξαχθούν και να ολοκληρωθούν κιόλα. Αυτά τα πειράματα, αυτή η έλεγχη, ώστε να συναυθεί και αυτή η συμφωνία τόσο σημαντική για τη Γεωργία. Πρόεδρο ευχαριστούμε. Σχέδιο έκθεση υπάρχει. Προθεσμία για την υποβολή του υπολογιών αύριο στι 6 το απόγευμα. Περνάμε στο σημείο 12. Εξυγχρονισμός των τελωνίων. Γνωμοδότηση της ΥΜΚΟ. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης που έχετε στα ντοσχέ σας. Η συγγήτριά μας, η κυρία Μουσκαρντίνη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε θα είμαι συνοπτική, διότι τα έχουμε συζητήσει και σε άλλες περιστάσεις στην Επιτροπή μας πανελειμμένως. Και ακριβώς με την παρουσία του Επιτρόπου Ντεχούχτ. Εδώ απλώς γνωματεύουμε ε, για την γνωμοδότηση της ΙΜΚΟ, όμως πρέπει εδώ να γίνει σαφές ότι για τα τελωνία που είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει, που είναι εργαλείο προστασίας των καταναλωτών καταπολέμησης της ε, προσέλευσης, της έλευσης μάλλον παράνομων ή παραποιημένων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση <clears throat> εκεί υπάρχει ανάγκη εναρμόνισης στη διαχείριση των ε, τελωνίων. Ιδάλλως οι εθνικές αρμοδιότητες πλήττουν ε, την, με τον κατακαιρματισμό τους την ε, εμπορική δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα υπάρχουν διαφορετικά μέτρα και σταθμά ανάλογα με το τελειωνικό σύστημα που χρησιμοποιεί κάθε χώρα. Παράδειγμα, εμπορεύματα που σε κάποιες χώρες εκτελονίζονται με συγκεκριμένο ποσοστό ΦΠΑ, σε άλλες χώρες έχουν άλλο ποσοστό να επιβάλλεται. Προφανώ ο εξαγωγέα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση θα κοιτάξει να πάει εκεί που είναι χαμηλότερο ο ΦΠΑ. Ακόμη και αν ε, η πιο, ο πιο ακριβώ ΦΠΑ μπορεί να σημαίνει και λιγότερου ελέγχου. Ποια θα είναι η συνέπεια λοιπόν, θα προσφέρονται προϊόντα στους Ευρωπαίους καταναλωτές που μπήκαν με δασμολόγηση και σύστημα ελέγχου διαφορετικό. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει συνέπεια στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, καλούμε μάλλον την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να εναρμονίσουν περαιτέρω το τελωνιακό του σύστημα, ώστε να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει ομοιόμορφη υλοποίηση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προστασία των καταναλωτών, σεβασμός των καταναλωτών. Για την ισορροπία της έκθεσης αυτής, βεβαίως, ζητούμε και μεγαλύτερη εύνοια για το εμπόριο, ώστε να ελεγχθούν καλύτερα και πληρέστερα οι πολυμερείς συμφωνίες. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε ο κύριος Ανδρέας. Η κυρία Ανδρέας. Η κυρία Ανδρέας Βαρέα. Μιλά εκ μέρους του Λούκα Σούστα που δεν είναι εδώ. Και θα διαβάσω αυτά ακριβώς που μου άφησε. Και θα ξεκινήσω λέγοντας, ζητά γνώμη για την απουσία μου. Ευχαριστώ την εισηγήτρια μου Σκαρδίνη για την έκθεσή της που υποβάλλεται σήμερα. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για το οποίο ζητήθηκε γνωμοδότηση από την πλευρά μας όσον αφορά την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτών. Υπάρχει ο κώδικας των τελωνίων ο οποίος ε, δυστυχώς όμως δεν είναι έτοιμος, ναι, διακόπτει ο πρόεδρος. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να μεταφραστεί έτσι γρήγορα όπως διαβάζετε. Πιο αργά παρακαλώ, για να μπορούν να σας μεταφράσουν και οι διερμηνείς. Τα πρόσφατα χρόνια διαπιστώσαμε μια σημαντική αύξηση του όγκου του διεθνούς εμπορίου, κάτι το οποίο οδήγησε τα τελωνία να αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι πολύ βασικό να διασφαλίσετε η ασφάλεια στα σύνορα, να προστατεύονται οι καταναλωτές και να προστατεύονται και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όσον αφορά το σχέδιο γνωμοδότηση, συμφωνώ απόλυτα με το μεγαλύτερο μέρος των ιδεών και των προτάσεων της εισηγήτριας. Πρέπει πράγματι να έχουμε τελωνία όλο και πιο αποτελεσματικά. Είναι απαραίτητο να μειώσουμε τον αριθμό των διαδικασιών των περιτών Συγχρόνως όμως πρέπει να ενισχυθεί το επίπεδο ασφάλειας. Πρέπει να τυποποιηθούν οι προδιαγραφές και η νομοθεσία των διαφόρων χωρών έτσι ώστε να έχουμε την ίδια ποιότητα ελέγχου μεταξύ όλων των κρατών χωρών και δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης και τον εξυγχρονισμό των διαδικασιών που να συνάδουν με τα τεχνολογικά επιτεύγματα. Χρειάζεται βέβαια, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη επένδυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Η διεθνή συνεργασία στον τομέα αυτό είναι κάτι που πρέπει να προωθηθεί και γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε τη διμερή συνεργασία με τους κύριους εμπορικούς μας εταίρους και επιπλέον να δουλέψουμε πιο δραστήρια και στο πολυμερές επίπεδο με τον ΠΟΕ και την ε, Παγκόσμια Οργάνωση Τελωνίων. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για όλες τις διεθνείς συναλλαγές. Ευχαρίστως να συνεργαστώ και με την εισηγήτρια και με τους άλλους σκιώδες εισηγητές έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα κοινό κείμενο από τη δικιά μας Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σιλβάνα Κοχαμέριν έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την ε, πληρέστατη αυτή γνωμοδότηση. Λίγα έχω να προσθέσω δύο μόνο στοιχεία που μπορώ να τα περάσω, αν μπορέσω και μέσα από τροπολογίες. Καταρχήν, η κατάργηση των προφορικών τελωνιακών δηλώσεων που ισχύει σε κάποια κράτη, δεν το προβλέπει το σχέδιο της Κομισιόν πλέον αυτό, είναι σημαντικό υπήρξε ανταλλαγή επιστολών μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το θέμα και της Επιτροπής ΙΜΚΟ και τα παραδείγματα που αναφέρονται στην επιστολή του κυρίου Τζεμέτα δεν ήταν τόσο πιστικά γιατί αναφέρονταν σε ιδιωτικές εισαγωγές και όχι ε, βιομηχανικές. Και η αιτιολόγηση ε, δεν ήταν σωστή για την κατάργηση της ε, προφορικής δήλωσης. Εμείς πρέπει να τη διατηρήσουμε αυτή τη μέθοδο νομίζω. Αυτό ήταν ένα που ήθελα να τονίσω και το άλλο αφορά πάλι ένα θέμα που συζητήθηκε, δηλαδή η εισαγωγή κανόνων για τους καταλόγους όπου πρόκειται ας πούμε για την καταγωγή του προϊόντος, κανόνες προέλευσης Υπάρχει μια συμβιβαστική λύση η οποία τώρα αμφισβητείται από το σχέδιο της Κομισιόν. Και θα πρέπει να δούμε το ζήτημα με ιδιαίτερη προσοχή. Δεν μας ευχαριστούν όλα όσα συμβαίνουν στην περίπτωση αυτή. Θα προβάλλουμε λοιπόν τροπολογία σχετικά ώστε να επιληθεί το ζήτημα και να ληφθεί υπόψη από τον εισηγητή. Ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Ραβέ από την Ταξούντ. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνεται στην εισηγήτρια και την Επιτροπή σας, όχι για πρώτη φορά, για την έκθεση αυτή εξυγχρονισμού των τελωνίων στην ενιαία αγορά. Και βλέπουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι οι βουλευτέ τη Επιτροπή σα αναγνωρίζουν τον καθοριστικό ρόλο των τελωνίων στην προστασία τη κοινωνία, αλλά και τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου. Αυτά είναι καθοριστικοί παράγοντε της οικονομική ανάπτυξη. Όπω είπε και η τα τελωνία όλο και περισσότερο εφαρμόζουν μέτρα στο επίπεδο των συνόρων για να αναχαιτήσουν κινδύνους για την ασφάλεια, την προστασία και το περιβάλλον. Τα τελωνία διδραματίζουν ένα κέριο ρόλο και για την ευρωπαϊκή οικονομία, όπω με την υλοποίηση, όπω υπόθηκε, για τα δικαιώματα πνευματική και δυνατική ιδιοκτησία. Ε, έχουν λοιπόν ε, την ε, αρμοδιότητα και την δυνατότητα τα τελωνία να φέρουν ει πέρα τέτοιο ρόλο, όπω έχουν αποδείξει ω τώρα εμπορικέ ροέ. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φροντίζει να εξυγχρονίσει την νομοθεσία τη, ώστε να δώσει ένα περιβάλλον διαλειτουργικό για την καλή λειτουργία των τελωνίων, για τον εξυγχρονισμό του κώδικα που, τους, που τα διέπει και για την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων με τα τελωνία. Όπως υπόθηκε, δεν είναι ακόμη το σύστημα πλήρως ενδρομονισμένο, ούτε ολοκληρωμένο, και το Κοινοβούλιο απίθυνε έκκληση μέσω του Προέδρου της Επιτροπής ΙΝΤΑ. Ίσως να υπάρξει αναβολή του συλλοποίηση, του τελευταίου, του πιο πρόσφατου κώδικα τελωνιακού, όμως θα πρέπει ήδη να αρχίσουμε να αντλούμε ωφέλη από αυτή τη διαδικασία εξυγχρονισμού. Επειδή θα είναι πολλέ οι των τελωνίων, πρέπει να δούμε και πιο συγκεκριμένα σημεία, όπω αναφέρονται στην έκθεση σε σχέση με το ευρωπαϊκό καθεστώς, τους δασμούς και τα όσα γίνονται στον τομέα της διαχείρισης των κινδύνων των τελωνιακών ελέγχων, τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και των τελωνιακών κυρώσεων. Αρκετοί βουλευτές αναφέρθηκαν στο τι γίνεται με το ΦΠΑ κατά τις εισαγωγές ή τις βιώσιμες ε, τελωνιακές δηλώσεις, αν καλά το κατάλαβα, αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά, ιδίως για το τελευταίο σημείο. Πολλές επαφές υπήρξαν μεταξύ βουλευτών και επιτροπής γι' αυτό. Και ελπίζουμε ότι θα βρούμε μια λύση που ικανοποιεί και τις απαιτήσεις για λιγότερη χρήση χάρτου και για να αντλήσουμε και περισσότερα ωφέλη. Σε όλους αυτούς τους τομείς χρειαζόμαστε τη στήριξή σας για να εξεύρουμε την ορθή ισορροπία μεταξύ της απαραίτητου επίπεδου προστασίας και της νόμιμης διευκόλυνσης του εμπορίου. Ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Mm, Ευχαριστώ. Τελευταίες παρατηρήσεις. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Οι τροπολογίες πιστεύω ότι θα βελτιώσουν την έκθεση. Απλώς να θυμίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξή. Για ένα θέμα τόσο κατεπήγον, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αναβάλουμε την εξετασή του. Πρέπει να αρχίσουμε να οδεύουμε προς την ολοκλήρωση τα τελωνία. Βρίσκονται στα εξωτερικά μας σύνορα. Είναι η μόνη μας εγγύηση, η μόνη μας διασφάλιση για να αποφύγουμε παραποιημένα ή παράνομα εμπόρια να φτάνουν στην επικράτεια της Ένωσης. Αν έχουμε διαφορετικά συστήματα, διαφορετικά ωράρια στη λειτουργία των τελωνίων και διαφορετικό κόστος, είναι προφανές ότι δεν θα είμαστε σε θέση σε όλου του Ευρωπαίου πολίτε να διασφαλίσουμε τι ίδιε εγγύσει, το ίδιο επίπεδο προστασία. Γι' αυτό τα τελωνία πρέπει να ενοποιηθούν. Εάν η εσωτερική αγορά θέλουμε να λειτουργεί σωστά και εύρυθμα. Εάν ξεκινούμε από τη λογική ότι η ευρωπαϊκή αγορά θα λειτουργεί όπω να είναι, α παρατήσουμε τα τελωνία στην τύχη του. Και το διεθνέ εμπόριο α, έχει διαφορετικού κανόνε ανάλογα με το ποιο σύνορο θέλει να περάσει. Από ποιο σύνορο θέλει να περάσει το εμπόρευμα. Ευχαριστούμε προς θεσμία για την υποβολή των τροπολογιών αύριο στις 6 το απόγευμα. Όπως προγραμματίζεται η οθέτηση της έκθεσης στην Επιτροπή μας 11 Οκτωβρίου. Και περνάμε στο επόμενο σημείο 13. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και τα αλληλευτικά προϊόντα. Σήμερα θα έχουμε τη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων με συμμετοχή εξωτερικών ε, προσκεκλημένων. Τον Ιούλιο συζητήσαμε πρώτη φορά με τους πολιτικούς συθήνοντες και για σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδρέας Γκόγκορα, είναι προσωρινός γραμματέας της συντονίστριας των γεωργικών προϊόντων και κτηνοτρόφων της Ισπανίας, ο κύριος Ζορ Ζουρντό, γενικός διευθυντής του, της αγοράς Σανσάλ, Περπινιό και Φόνς, η κυρία Ανζελίκ Ντελαχέ, πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Εμπόρων Οπροκυπευτικών, και ο κύριος Μανφρέντο Φάντι, από, την, από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ο κύριος Νίκολας Ελέα από την Γενική Διεύθυνση Άγκρη, που είναι, και πρόεδρος, που είναι πρόεδροι μάλλον και αντιπρόεδροι αντιστοίχως, της Επιτροπής Γεωργικών Προϊόντων και Αλληλείας της, της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου βρίσκονται εδώ γιατί η Επιτροπή του παρακολουθεί το πώ θα τεθεί σε ισχύ η συμφωνία και ο κύριο Φάντη καθώ ο κύριο Ελέ είναι πρόθυμοι να συζητήσουν με τα μέλη τη Επιτροπή για το πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διασφαλίσει την ορθή ολοποίηση τη ε, συμφωνία αυτή. Έχουμε επίση τον κύριο Τζον Κλάρκ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπεύθυνο για τι διεθνεί σχέσει τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη. Α ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω. να δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας. Πέντε λεπτά στον καθένα. Μετά θα δω, πάρουν το λόγο οι βουλευτές, με κύριο Σοφάντα και ο κύριος Βερλέ και τέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά και ο εισηγητής μας για τις καταληκτικές παρατηρήσεις. Το ζήτημα θα το ολοκληρώσουμε Αποφασίζοντα με τις ημερομηνίε τι θα γίνει, γιατί ακόμα δεν υπάρχει σχετική απόφαση. Α ξεκινήσουμε με την ε, παρουσίαση του κυρίου Γκόγκορα. Ισπανό Ισπανός ε, ο κύριος Γκόγκορα, όπως είπα, από το συντονιστικό όργανο γεωργών και Εκτινοτρόφων. Sí, hola. Muy buenas tardes a todos. Eh, mi nombre es Andrés Ευχαριστώ. Είμαι υπεύθυνο του τμήματο οποροκυπευτικών του επαγγελματικού κλάδου της Ισπανίας. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ την Επιτροπή σας που μας προσκάλεσε να έρθουμε εδώ και να συμμετάσχουμε στην ανταλλαγή απόψεων. Ελπίζω η παρέμβασή μου να αποβεί χρήσιμη για την εφαρμογή ορθών μέτρων όσον αφορά το θέμα μας. Είμαι και εγώ αγρότης. Ζω στην Αλμερία, στην νοτιοανατολική ε, Ισπανία και είμαι τρίτη γενιά ο Γεωργού εκεί στην περιοχή με τα παροκυπευτικά που ασχολούμαι. Η κρίση πλήττει και τον δικό μας τον τομέα. Υποφέρει και γι' αυτό έχουμε πάρα πολλές αμφιβολίες κατά πόσο η συμφωνία αυτή είναι επωφελής για μας. Στο λίγο χρόνο που έχω στη διαθεσή μου θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω γιατί αποτελεί ένα βαρύ χτύπημα στη σποδηλική στήλη των οποροκυπευτικών της Μεσογείου. Δεν προσφέρει τίποτα ούτε στους Ευρωπαίους καταναλωτές, ούτε και στους ε, Σαραουί που κι αυτοί είναι παραγωγή οποροκυπευτικών και που θα έπρεπε να μπορούν να επωφεληθούν από την ε, συμφωνία αυτή ελευθέρωσης. Το θέμα που συζητιέται σήμερα, η ανανέωση της συμφωνής αυτής, δεν αφορά την ντομάτα, όπως λέμε συχνά, αλλά πρόκειται για την ελευθέρωση ουσιαστικά ολόκληρου του τομέα απορροκυπευτικών από το Μαρόκο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντα μιλάμε για την ντομάτα, ενώ στην πραγματικότητα δεν πρόκειται μόνο για την ντομάτα. Θα θέλαμε επίσης να σας δώσουμε και κάποια στοιχεία συγκεκριμένα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε σημείο αναφοράς για να καταλάβετε περί τίνος μιλάμε όταν μιλάμε για τα ποροκυπευτικά στην Ευρώπη. Είμαστε το 3% της καλλιεργήσιμης γης στην Ευρώπη. Έχουμε όμως 1.400.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο, μεγάλο πόσο πολύ εργατικό δυναμικό απασχολείται στον τομέα αυτό. 17% της γεωργικής ευρωπαϊκής παραγωγής, πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Και άρα είμαστε ο πιο σημαντικός τομέας από όλους τους γεωργικούς και κτηνοτροφικούς τομείς, είτε πρόκειται για δημητριακά, είτε για γάλα, είτε για άλλους ε, τομείς. Δημιουργούμε θέσεις απασχόλησης και άμεσα, μια που σας είπα ότι πρόκειται για 1.400.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και έμεσα, διότι οι εκμεταλλεύσεις αυτές με τη σειρά τους δίνουν δουλειά σε άλλους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε. Στην Ισπανία, εκεί από όπου προέρχομαι εγώ, ο τομέας αυτός προκυπευτικών έχει τεράστια σημασία. 14 εκατομμύρια και κάτι πολύ σημαντικό σε σχέση με τη συνολική παραγωγή. Και είναι μάλιστα ένα τομέας ο οποίος δεν παίρνει ενισχύσεις από την ΚΑΠ, μόνο 3% ολόκληρου του όγκου χρημάτων που δίνεται στην ΚΑΠ, μόνο το 3% παίρνουμε εμείς. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι τα έσοδά μας έρχονται πραγματικά από την παραγωγή. Παρ' όλα αυτά, είμαστε το 40% απασχόλησης ε, στη γεωργία ε, μέσα σε ολόκληρη την Ισπανία. Που σημαίνει ότι ζούμε από την αγορά. Δηλαδή οποιοδήποτε άνοιγμα εμπορικό οδηγεί σε αποσταθεροποίηση της εσωτερικής αγοράς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σημαίνει μεγάλο χτύπημα στην αποδοτικότητα και μπαίνει σε κίνδυνο η απασχόληση της γενιάς αυτής. Γι' αυτό λοιπόν και ζητάμε να έχετε υπόψη σας τα στοιχεία αυτά, αλλά και άλλα τα οποία σας δίνω. Όπως έλεγα και πριν, εμείς καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει η γεωργία και καταλαβαίνουμε, σαν αγρότες που είμαστε, πόσο μεγάλη σημασία έχει να έχουμε εμπορικέ σχέσεις με την Βόρεια Αφρική, με το Μαρόκο. Σύμφωνοι. Είναι όμως πολύ σημαντικό ό,τι συμφωνίες κάνουμε μαζί τους να διασφαλίσουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας και το μέλλον των πολιτών της Βόρειας Αφρικής. Η συμφωνία αυτή λοιπόν δεν διασφαλίζει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Επιπλέον θέλω να υπογραμμίσω εδώ ότι όπως πολύ σωστά αναγνώρισε και η ίδια η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μελέτη αντικτύπου, οι επιπτώσεις από την εμπορική ελευθέρωση αυτή, δεν έχουμε την μελέτη αντικτύπου όσον αφορά την ε, συμφωνία με το Μαρόκο, αλλά από άλλες αντίστοιχες λέει ότι αυτοί που έχουν να περισσότερο είναι η παραγωγή οποροκυπευτικών. Γιατί δεν μπορούμε τότε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Είναι λοιπόν απαραίτητο να κοιτάξουμε αυτή η εμπορική ελευθέρωση του τομέα έχει κάποιο θετικό για τους Ευρωπαίους πολίτες ή για τους πολίτες της Δυτικής Αχάρας οι οποίοι τελικά βλέπουν την παραγωγή τους να περνάει από τα χέρια μεγάλων πολυεθνικών. Άρα δεν πρόκειται να υποφεληθούν οι ντόπιοι παραγωγοί, κάθε άλλο. Τα πλεονάσματα τελικά επαναδιανύμονται και κάνουν μεγαλύτερη ζημιά στους παραγωγούς. Ναι, ναι, τελειώνω. Η διαδικασία αυτή εμπορικής ελευθέρωσης δεν βοήθησε ούτε καν για ενίσχυση της δημοκρατίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων της περιοχής όπου βρίσκονται οι εκμεταλλεύσεις αυτές. Ευχαριστούμε πολύ, διακόπτει ο Πρόεδρος. Επόμενος. Ο κύριος Ζουρτώ. Γενικός Διευθυντής ο κύριος Ζορντών από το Περπινιό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι η Saint Charles International είναι το πιο σημαντικό κέντρο της Ευρώπης. Φτάνουν σε εμά προϊόντα τα οποία διανέμουμε στη Γαλλία και στην Ευρώπη. Η Saint Charles έχει δύο άξονες. Πρώτα απ' όλα τον Ισπανικό και έπειτα εκείνον του Μαρόκου αλλά και κάποιους άλλους πολύ πιο ασήμαντους. Αυτό που είναι σημαντικό να πούμε για τη συμφωνία αυτή που υποβάλλεται προς έγκριση στο Κοινοβούλιο είναι ότι η συμφωνία αυτή έχει να κάνει με το δικό καθεστώς ε, του Μαρόκου που είναι αρκετά προωθημένο και δεν βρίσκεται σε βαθμό πλήρης ελευθέρωσης. Όχι, είναι σε ένα βαθμό. Για μας λοιπόν η συμφωνία αυτή, η ελευθέρωση αυτή θα επιτρέψει στο σύνολο των ε, Ευρωπαίων εξαγωγών υποφεληθούν από την αγορά του Μαρόκο. Γιατί στον γεωργικό τομέα ξέρουμε ότι η ελευθέρωση του 45% όπως συμφωνήθηκε σε αξία και 70% σε 10 χρόνια. Υπάρχει βέβαια μια συμμετρία, όμως η συμφωνία αυτή είναι προτιμότερη από πλήρης άνοιγμα της ε, Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει ένα πραγματικό άνοιγμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με μια χώρα όπου η παραγωγή αλλάζει και όπου δημογραφικά υπάρχει τεράστια αύξηση. Υπάρχουν σημαντικές ε, παραχωρήσεις, γίνεται αύξηση και για τα δημητριακά και για τα ποροκυπευτικά και για το γάλα και για τα όσπρια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι η ευαισθητοποίηση του τομέα παροκυπευτικών έχει ληφθεί υπόψη. Οι ποσοστώσει οι δασμολογικέ έχουν διατηρηθεί για τα ευαίσθητα προϊόντα. Για την ντομάτα, η οποία διακυδεύεται ε, εδώ, περιορίστηκε η αύξηση για πέντε χρόνια με μια διατήρηση ε, τελών η επίσης αρχή της συμπληρωματικότητας των παραγωγών εκατέρωθων της Μεσογείου είναι κάτι που επίσης διατηρήσαμε, όπως επίσης διατηρήθηκε και το καθεστώς της τιμής εισόδου. Ο σεβασμός των διεθνών συμφωνιών επίσης για τα υγειονομικά και φυτογειονομικά πρότυπα είναι κάτι που επίσης διατηρείται και τηρείται. Οπότε σε σχέση με τη σημερινή συμφωνία πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το εμπορικό ισοζύγιο σήμερα ανάμεσα στο Μαρόκο και την Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοεί τους Ευρωπαίους. 12,7 δις προϊόντα ενώ 7,3 δισεκατομμύρια είναι οι εισαγωγές. Στο 1,2 εκατομμύρια τόνους, γιατί βέβαια μιλάμε για τα πορκυπευτικά εδώ, 850.000 τόνοι τυχαίων επεξεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1 τρίτο ντομάτα. Εμείς είμαστε 75% των όσων ε, ξεργαζόμαστε σε επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν αντικειμενικά σήμερα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία αύξηση της κυκλοφορίας το βλέπουμε αυτό εμείς, ιδιαίτερα για την Ισπανία. Κατά μέσο όρο τα τελευταία τρία χρόνια είχαμε αύξηση 20% της κυκλοφορίας, αλλά έχουμε λιγότερη αύξηση 4% όσον αφορά τα φρούτα από το Μαρόκο. Πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι αντίθετα με αυτό που λέγεται δεν επωφελούνται οι μεγάλες εταιρείε του Μαρόκο, όχι, αλλά οι μικροί συνεταιρισμοί οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν βάζοντας μαζί τα λογιστικά τους μέσα. Τώρα για τις αγωγές, πέρα από τη δουλειά που έχει γίνει από την Επιτροπή, πρέπει να σας πούμε εδώ, έχοντας διασταυρώσει πληροφορίες, ότι εμείς έχουμε μια βάση δεδομένων μοναδική στην Ευρώπη, η οποία μας επιτρέπει ε, να γνωρίζουμε ακριβώς τις εμπορικές ροές. Επίσης και όσον αφορά την εποπτεία των εισαγωγών, μπορούμε εδώ να πούμε ότι σήμερα δεν υπάρχει καμία υπέρβαση των δασμολογικών ποσοστώσεων. Αντίθετα, είναι σαφές και το ξέρουν όλοι, το Μαρόκο μπορεί στα πλαίσια των συμφωνιών που έχει στον ΠΟΕ να ξεπεράσει τις συμφωνίες αυτές με τα προϊόντα του. Όσον αφορά τώρα την τιμή εισόδου, πρέπει να ξέρουμε ότι η τιμή αυτή ρυθμίζει την κατάσταση. Από τη στιγμή που εκαθαδρύθηκε, σταθεροποιήθηκε η αγορά. Στη συνέχεια, ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η υγειονομική και η φυτογειονομική ρύθμιση. Εδώ πρέπει να ξέρουμε ότι από τις έρευνες που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν ότι δεν έχουμε περισσότερες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης από το Μαρόκο σε σχέση με άλλα προϊόντα που μας έρχονται από τρίτες χώρες ή από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Εμείς στη Σανσάρλ έχουμε φροντίσει να εξετάζουμε την ποιότητα και εμείς φροντίζουμε κάθε φορά όταν υπάρχει ε, χαμηλότερη ποιότητα να φροντίσουμε να απορρίπτουμε. Και έτσι διατηρείται μια ποιότητα ίδια με εκείνη που έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να επιμείνω στο εξή. Έχουμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη κρίση. Και να υπενθυμίσω ότι να τα βάζουμε, ιδίως επειδή είχαμε την κρίση με το e να τα βάζουμε με, τη, με ένα συγκεκριμένο προϊόν είναι σαν να τα βάζουμε τον καταναλωτή. Πρέπει να δώσουμε νέο δυναμισμό στον τομέα μας και να φροντίσουμε τα προϊόντα μας να καταναλώνονται εν ασφαλεία και χωρίς κανένα κίνδυνο. Ευχαριστώ. Τέλος, η κυρία Ντέλα Ε, πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Εμπόρων Προκυπευτικών. Ε, ε, ε, α, Και εσείς πέντε λεπτά. Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που μας προσκαλέσατε και οργανώσατε αυτή τη συζήτηση σε σχέση με την ε, Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου. Βεβαίως, δεν θα επαναλάβω τα όσα είπε ο Ισπανός συνάδελφος. Συμφωνώ απολύτως. Απλώς θέλω να επικεντρωθώ σε έναν τομέα παραγωγής, πολύ σημαντικό για τη Γαλλία, της ντομάτας. Σήμερα ε, είναι αυτό ο τομέας που περισσότερο πλήττεται από την αναθεώρηση της ε, Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωση Μαρόκου. Να πω απλώς ότι η ντομάτα είναι το πρώτο προϊόν που εξάγεται προ τη Γαλλία από την κατηγορία των οφοροκυπευτικών και βεβαίω υπάρχει επίδραση και στους υπόλοιπους τομείς ε, τροφίμων. Για την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεγάλο μέρος της ντομάτας που καταναλώνεται στη Γαλλία προέρχεται από το Μαρόκο. Άρα μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος να παραμείνει ισόρροπη αγορά στην επικράτειά μας, ιδίως ως προς την παραγωγή ντομάτας θερμοκηπίου. Αυτό που θέλουμε σήμερα να σας καταστήσουμε σαφές είναι σε πόσο μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας διαταράσει την ισορροπία των αγορών μας. Ιδιαιτέρως έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια μέσω των προηγούμενων συμφωνιών και την ε, θέση σε ισχύ τους ότι η τιμή έχει βελτιωθεί και έχουμε υπερβεί τα όρια των ε, ποσοτήτων που είχαν ε, αποδοθεί στο Μαρόκο. Μπορώ να σας δώσω κάποια στοιχεία για να στηρίξω τα λεγόμενά μου, καθώς και για τη ρήτρα διασφάλισης να πω ότι φάνηκε να είναι τελείω αναποτελεσματική. Δεν χρησιμεύσε σε τίποτα. Κατά τα άλλα θέλω να υπογραμμίσω ότι ο τομέας αυτός είναι σημαντικός για ολόκληρη την Ευρώπη η παραγωγή στο θερμοκηπίου. 40.000 θέσεις εργασίας στη Γαλλία, αμέσως και αμέσως. Ακόμη και για μη τυποποιημένες επαγγελματικές θέσεις. Η επίδραση λοιπόν της συμφωνίας αυτής μέσω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης στην Ευρώπη θα μας πλήξει ιδιαίτερος. Μας φαίνεται σημαντικό προτού υπογραφεί οποιαδήποτε συμφωνία να υπάρξει μελέτη αντικτύπου για το κοινωνικό και το οικονομικό επίπεδο στις ζώνες παραγωγής ντομάτας θερμοκηπίου ιδιαίτερος. Το θερμοκήπιο για την παραγωγή των λαχανικών είναι ένας από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς και τους πλέον ζωντανούς. Είναι ένα εργαλείο που επέτρεψε την ε, βελτίωση κάποιων ε, στοιχείων της παραγωγής, ιδίως την, ε, τις καλές συνθήκες εργασίας, κάτι που σπανίως αναπτύσσετε στι συζητήσει που θίγουν τα γεωργικά ζητήματα, διότι σήμερα η γεωργία πραγματικά προσφέρει θέσεις εργασία που επιτρέπει στου εργαζόμενους να εργάζονται σε αξιοπρεπείς συνθήκε, δεδομένου και του κοινωνικού πλαισίου εντό του οποίου ζούμε. Μπορούμε έτσι να διατηρήσουμε και έναν δυναμικό γεωργικό ιστό και χάρη σε όλα αυτά να αναπτύσσονται άξονες όπως το δίκτυο του φυσικού αερίου Χωρίς την ύπαρξη των θερμοκηπίων και των υπευθύνων τους, δεν θα ήταν αρκετά αναπτυγμένο σε εθνικό επίπεδο. Άλλα σημεία που τα θεωρούμε σημαντικά είναι η τιμή εισόδου. Η εισαγωγή ενός κιλού ντομάτα στην Ευρώπη σημαίνει μεταφορά 100 λίτρων νερού. Η παραγωγή στην Ευρώπη ενός κιλού στην ε, Ευρώπη σημαίνει κατανάλωση 12,5 λίτρων νερού. Μπορούμε να επιτρέψουμε στο εαυτού μα να αποξηράνουν τελείω χώρε όπω το Μαρόκο, ενώ εμείς εδώ έχουμε πολύ χαμηλότερη κατανάλωση, ιδίω στην Ευρώπη. Χάρη στα θερμοκήπια έχουν γίνει σημαντικές εξοικονομήσεις ενέργειας επίσης. Σήμερα πολλέ από τις εγκαταστάσεις μας λειτουργούν με βιομάζα ή με τη συμπαραγωγή όπως λέγεται παράδειγμα το τι συμβαίνει στις κάτω χώρες με τα θερμοκήπια. Σήμερα το θερμοκήπιο γίνεται εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού πριν γίνει εργοστάσιο λαχανικών. Επίσης και ως προς τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα είναι πολύ αποτελεσματικά τα θερμοκήπια. Νομίζω αυτή είναι μια από τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη τα ερχόμενα χρόνια. Και για όσους λένε ότι οι εισαγωγές δεν είναι, μάλλον υποστηρίζουμε και εμείς ότι οι εισαγωγές δεν είναι καθαρή περιβαλλοντική λύση. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που ήδη ισχύουν πολύ συχνά παρακάμπτονται. Πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά προηγουμένως ε, πώς θα διοργανωθεί όλο αυτό το σύστημα προκειμένου να καταρτιστεί σωστά η νέα συμφωνία. Ε, η τιμή εισόδου θα πρέπει να λειτουργεί ανάλογα με το πώς ε, κατανέμεται το προϊόν και για να μην υπάρξει κοινωνικό dumping. Χωρίς αυτού του είδους τον προηγούμενο προβληματισμό, η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών όπως προβλέπετε θα αποσταθεροποιήσει μόνιμα έναν τομέα που ήδη βρίσκεται σε κρίση. Θα καταστραφούν όλες οι προσπάθειες των Γάλλων και Ευρωπαίων παραγωγών προκειμένου να διοργανωθούν σε αυτόν τον τομέα παραγωγής. Είναι λοιπόν ε, απαραίτητο να σκεφτείτε προσεκτικά την, ε, το σχεδιασμό αυτής της συμφωνίας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις σας. Προχωρούμε στη συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής μας. Ξεκινούμε με τους σκιώδεις εισηγητές. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε χρόνο. Περιορισμός λοιπόν. Δύο λεπτά για τον καθένα. Έχω πάρα πολλούς ε, αγορητές. Ο κύριος Γιακολίνο από το ΕΛΚ. Πρόεδρε, άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τις παρεμβάσεις των προσκεκλημένων μας και των ε, θετικών και των αρνητικών ως προς τη συμφωνία. Προφανώς, οποιαδήποτε συμφωνία προκαλεί προβληματισμό σε κάθε περίπτωση υπάρχει ήδη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου ακριβώς για τα συγκεκριμένα ζητήματα που σήμερα θίγησαν. Η πολιτική για την Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει προφανώς το σεβασμό προς το Μαρόκο που κατάφερε να εξασφαλίσει ατομικές ελευθερίες στους πολίτες του, τη δικαιοσύνη, την απαραίτητη ισορροπία που επέτρεψε να αποφευχθούν φαινόμενα όπως αυτά που γνώρισαν οι άλλες χώρες της Βορειοαφρικής. Η συνεργασία του Ευρωκοινοβουλίου και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων είναι απαραίτητη. Θα ενισχύσουν την πνοή ελευθερίας και ειρήνης που μας έρχεται από το βασίλειο του Μαρόκου. Επίσης, το Μαρόκο έχει πάντοτε πολύ ε, αρμονικές σχέσεις μαζί μας. Βεβαίω, στη χώρα υπάρχουν και κάποιε πραγματικότητες που ε, μας επιτρέπουν να κάνουμε κι εμείς κάποιες παρατηρήσεις. Τα οποροκυπευτικά και η ντομάτα μπορεί να πληγούν από μια συμφωνία που θα απελευθερώσει την εμπορία πολλών προϊόντων. Θα υπάρχουν διαφορές στην επιβολή δασμών. Θα υπάρχει δυσκολία με την ε, γεωγραφική χνηλασιμότητα και την επισητιστική ασφάλεια, τις γεωγραφικές ενδείξεις των προϊόντων. Υπάρχουν ακόμη ενδιασμοί για τις θετικές ε, επιδράσεις και για τις διακυμάνσεις των τιμών, στη σημεία που έθιξαν η Επιτροπή Άγκρη και ΠΕΣ. οι ποσοστώσει που δεν γίνονται πάντοτε σεβαστές. Όλα αυτά ακούστηκαν, αλλά και η ρήτρα διασφάλιση. Πρέπει λοιπόν το θέμα να μελετηθεί περαιτέρω. Και μια γρήγορη ερώτηση προς την Επιτροπή. Ποιος θα είναι ο οικονομικός αντίκτυπος, τι θα αλλάξει ως προς την οικονομική αξία αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστούμε. Μαρία Αντσαρνές, την Άλντε. Ευχαριστώ. Ε, βρήκα τις παρουσιάσεις αυτές ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, διότι επί της ουσίας δεν έχουμε καταλήξει μια ενιαία θέση για τη συμφωνία αυτή. Εφόσον λοιπόν υπάρχει συζήτηση και αποκλήσεις της απόψεις, νομίζω ότι πλέον εναπόκειται σε εμά τους ευρωβουλευτές να εμβαθύνουμε στα ζητήματα. Εμένα η συμφωνία όπως μας παρουσιάζεται σήμερα δεν με ικανοποιεί. Η συμφωνία ε, πρέπει να αναρωτηθούμε αν είναι καλή για τους ε, Μαροκινούς, τους Αραουί ή τους Ευρωπαίου, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ναι σε καμία από αυτέ τι ερωτήσει. Έπειτα για αυτό το είδο συμφωνία. Πρέπει να αναρωτηθούμε για τι αρχέ μα. Ε, εμπορική ανάπτυξη ω αυτό σκοπό. Δεν νομίζω ότι αρκεί αυτό για μια χώρα. Η τοπική παραγωγή αναζητούν τη βιωσιμότητα και την ε, σταθερότητα κι αυτή. Αυτό θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητά μα και όχι μόνο η εμπορική μέρημνα. Για το Μαρόκο λοιπόν η γεωργική ανάπτυξη δεν πρέπει να γίνει απλώς με σκοπό τις εξαγωγές ε, για μία κατηγορία προϊόντων. Θα πρέπει να δούμε τις ανάγκες των τοπικών παραγωγών. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Τρίτη παρατήρηση. Το είπατε προλίγου. Προφανώς θέλουμε να υπάρχει αμοιβαιότητα στις προδιαγραφές. Υπάρχει αυτή τη στιγμή τεράστια απόκληση ως προς το κόστος εργασίας προφανώς, αλλά και των περιβαλλοντικών, θητικών και φυτο-υγειονομικών προτύπων και για τους κανόνες προέλευσης. Δεν έχουν ακόμη οριστεί σωστά. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε μια θετική προσέγγιση προς το Μαρόκο, να βοηθήσουμε τους Μαροκινούς, διότι η Αραβική Άνοιξη μας ε, υποχρεώνει να έχουμε μια εταιρική σχέση πιο καρποφορά, θα πρέπει τη συμφωνία να τη δούμε από το φως των μελετών αντικτύπου. Να μην αποθαρρυνθεί το Μαρόκο, να συζητήσουμε. Αλλά να συζητήσουμε σε διαφορετικές βάσεις και να ορίσουμε αρχές και σκοπούς τους οποίους θέλουμε να καταλήξουμε, αλλά όχι με μόνο σκοπό την ελεύθερη, τις ελεύθερες συναλλαγές ε, και με μόνο ε, να ωφελείται το εμπόριο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Βλέπουμε ότι έχουμε εδώ Γάλλους και ισπανού εκπροσώπους του γεωργικού τομέα. Είναι σημαντικό να τους ακούσουμε και να αναλύσουμε τόσα μα είπαν. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα λάβουμε υπόψη μα τις θέσεις τους και θα δράσουμε ανάλογα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας και την άποψη της Επιτροπής Γεωργίας όσον αφορά τη συμφωνία αυτή. Τώρα θα σας μεταφέρω διάφορες σκέψεις μου. Πρώτον, ότι το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα είναι εντελώς διαφορετικό από το πλαίσιο εκείνο μέσα στο οποίο το 2009 προεχνηθήκαμε αυτή τη συμφωνία. Τότε η Ευρώπη και η Ισπανία ήταν αλλιώ. Σήμερα είναι σε πολύ πιο τραγική κατάσταση και ο τομέα σήμερα βρίσκεται σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ότι η οικονομία γενικά. Και η κατάσταση στο Μαρόκο επίσης έχει αλλάξει πολύ αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχουν αρκετοί μηχανισμοί ελέγχου ή εργαλεία τα οποία να μας επιτρέπουν να εποπτεύουμε την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής και από τις δύο πλευρές. Και θα ήθελα να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι πιστεύει γι' αυτό. Αλλά μην πιστεύετε ότι είμαστε κατά των εμπορικών συμφωνιών και αυτή τη συγκεκριμένη. Όχι, είμαστε υπέρ τη ενίσχυση του εμπορίου, αλλά είμαστε υπέρ ε, ενίσχυση ενό εμπορίου με ισορροπία, από την οποία συμφωνία να υποφελούνται και οι δύο πλευρέ και η Ευρώπη, η Ισπανία ιδιαίτερα, αλλά και το Μαρόκο, μην αμφιβάλλετε γι' αυτό. Είμαστε επίση υπέρ συμφωνιών που να είναι αμοιβέ που να διασφαλίσουν την τήρηση κάποιων ελάχιστων κοινωνικών προδιαγραφών, κάποιων ελάχιστων περιβαλλοντικών προδιαγραφών και πολύ σημαντικό πρέπει να υπάρχουν και υγειονομικές και φυτογειονομικές προδιαγραφές. Πρέπει να διασφαλίσουμε την ε, διάθεση τροφίμων, κάτι το οποίο δεν είναι τόσο εγκυμένο όπως νομίζαμε κάποτε. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν αναρωτιέμαι η συμφωνία αυτή εγγυάται για την εφαρμογή όλων αυτών των προποθέσεων. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρόεδρος ευχαριστούμε. Ο Χωσέφ Αντρές. Ή Χωσέφ Ευχαριστώ. Είναι η τελευταία συμφωνία που έχουμε με το Μαρόκο. Έχουμε ακούσει διάφορες παραβάσεις και ευχαριστώ πολύ όλους όσοι πήραν το λόγο για τόσα μας είπαν. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον πρώτο που πήρε το λόγο, αλλά εδώ να διαφοροποιηθώ λίγο. Κατάλαβα αυτά που μας είπε, ότι ναι, θέλει μια συμφωνία, αλλά μια συμφωνία με εγγύσεις. Ο δεύτερος που πήρε το λόγο, θέλω να ρωτήσω, γίνεται έλεγχος των ποσοστώσεων εισαγωγής στο Περπινιάν και αν ο έλεγχος αυτός γίνεται πλήρως και μαζί με τις ποσοστώσεις να ελέγχουν και την ποιότητα της τομάτας που μπαίνει με χαμηλούς δεσμούς. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι η κατάσταση στο Μαρόκο είναι ιδιαίτερη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μαρόκο χρειάζεται κάποιες αποχρώσεις Πάντως είναι βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη εκδοχή. Και γιατί. Πρώτον, για τη βάση της ποσοστώσης ιδιαίτερα στα ευαίσθητα προϊόντα μας, ιδιαίτερα την ντομάτα, στην οποία αναφερθήκαμε. Μιλάει επίσης για μια ρήτρα στη σελίδα 15 που λέει ότι εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά οι ρήτρες ασφαλείας, όχι μόνο εφόσον υπάρξει αύξηση του προϊόντος στην αγορά, αλλά επίσης εφόσον υπάρχουν και επιπτώσεις στον τομέα μεταποίησης. Υπάρχει μια διαφοροποίηση δηλαδή σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλα σημαντικά στοιχεία, όπως είναι η μη τήρηση της τιμής εισαγωγής, πράγμα το οποίο εμείς καταδικάζαμε πάντα, ότι πρέπει να υπάρξει τροποποίηση του κανονισμού όσον αφορά τις τιμές εισαγωγής ε, το έχουν αναγνωρίσει αυτό όλοι και επίσης εμείς πιστεύουμε ότι αυτό είναι ζωτική σημασία. Και όσον αφορά τις φυτογενομικές προδιαγραφές και εδώ πρέπει να είμαστε με ανοιχτά τα μάτια, να ελέγχουμε και το προϊόν αλλά και την προέλευσή του. Κάτι το οποίο γίνεται στην Ισπανία και στην Ευρώπη. Δεν γίνεται όμως στο Μαρόκο, γιατί δεν τηρεί τις προδιαγραφές του ΠΟΕ. Μιλήσαμε πριν για τα τελωνία και τους ελέγχους στα τελωνία. Πολύ σημαντικό και εδώ. Πρέπει να υπάρξει διόρθωση και έλεγχος. Η προηγούμενη έκθεση, εξάλλου, πολύ σωστά υπογραμμίζει το θέμα αυτό των τελωνίων και του ελέγχου που κάνουν ε, όσον αφορά το διεθνές εμπόριο. Ευχαριστούμε. Από την ΚΟΕ τώρα. Δύο λεπτά όμως, ε, ε κύριε Μέρφη. Συνήθως ξεπερνάτε το χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές για τις παρουσιάσεις. Εγώ θα έλεγα ότι οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μαρόκο είναι κλασικό παράδειγμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατικών δικαιωμάτων, όταν έρθουν σε επαφή και προσκρούσουν με μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όλα αυτά μπαίνουν στην άκρη. Κλασικό παράδειγμα οι αλληλευτικές συμφωνίες, νεοπικιοκρατικές σχεδόν, σε βάρος των ε, μαροκινών αλλιέων και του λαού της Δυτικής Σαχάρας. Ε, ξέρω ότι το έγγραφο της Κομισιόν τάσεται υπέρ της ε, συμφωνίας, αναφέροντας και την Αραβική Άνοιξη αν ψηφιστεί είναι κατά της Αραβικής Άνοιξης όμως. Δεν είναι πρώτη φορά που βλέπω το Κοινοβούλιο να προσπαθεί να ε, φέρει όλα αυτά τα δικαιώματα ε, κοντά στην ε, απελευθέρωση εμπορίου και συναλλαγών. Στην πραγματικότητα όμως θα πρέπει να ταχθούμε κατά της απελευθέρωσης αν βλάπτει τους μικρούς παραγωγούς. Το βασικό θέμα είναι η Δυτική Σαχάρα. Και πάλι είναι απίστευτο. Δόθηκαν διασφαλίσει στο Μαρόκο ότι η συμφωνία θα ωφελήσει τον τόπιο πληθυσμό και ότι έγιναν διαβουλεύσει σε περιφερειακό επίπεδο. Πολύ αστείο. Πρέπει να δεχτούμε δηλαδή τις διασφαλίσεις αυτέ. Ε, αυτή είναι η κυβέρνηση που αρνήθηκε την αυτοδιάθεση του λαού τη Δυτική Σαχάρα που δεν ε, κάνει ε, δημοψηφίσματα και δεν ακούει τα αποτελέσματα όταν γίνουν, ε, αγνοεί τις διαμαρτυρίες. Τι διασφαλίσεις λοιπόν έχουμε ότι θα ο κόσμος. Και ε, ρωτήθηκα λαό τη Δυτική Σαχάρα. Μπορούμε να έχουμε εκπροσώπου του λαού τη Δυτική Σαχάρα σε αυτέ τι συζητήσει. Ευχαριστώ. Τέλο η κυρία Μουσκαρντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οφείλω να πω ότι κάποιες συμπεριφορέ με κάνουν να αισθάνομαι σχιζοφρενής. Διότι τρέξαμε να εγκρίνουμε γρήγορα γρήγορα τις συμφωνίες με την Κορέα. Δεν λέμε όμως τίποτα από την άλλη για τις κινέζικες ντομάτες που μπορεί να είναι και δηλητηριασμένες και εισάγονται και παρανόμως και νόμιμα. Ενώ με το Μαρόκο είμαστε επανετυχοί σε μια συνεδρίαση που μου φαίνεται ότι αφορά κυρίως τους Γάλλους και τους Ισπανούς συναδέλφους και το λέω με κάθε φιλική διάθεση. Ε, κύριε Γκογκόρα, όταν μιλάτε για μεσογειακή γεωργία στο Μαρόκο, όσο και να δεν σας αρέσει, Μεσόγειος είναι και εκεί. Η ανάπτυξη των χωρών μας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας θα ευνοηθεί. Εάν στις άλλες χώρες που βρίσκονται στην απέναντι όχθη τους δώσουμε τη δυνατότητα και αυτές να αναπτυχθούν και να είναι εταίροι μας. Ιδάλλως θα πεινάσουμε όλοι. Και αγαπητέ κύριε Γάλμπα, πολύ σωστά λέτε ότι άλλαξε η κατάσταση σε σχέση με ε, την τελευταία τριετία. Εντάξει, σωστά, αλλά να σας ρωτήσω εγώ, ποιος φταίει, ε, το Μαρόκο ή οι δικές μας οι κυβερνήσεις κεντροαριστεράς και κεντροδεξιάς και τα θεσμικά μας όργανα που δεν ασχολήθηκαν με την ε, τραγωδία που λαμβάνει η χώρα στη Δυτική Σαχάρα. Ε, για μια παρατήρηση, το καλοκαίρι φέτο στο Πιατσεντίνο, που είναι μια από τι σημαντικότερε ε, ιταλικέ περιοχέ παραγωγή ντομάτα, γνωστή σε όλη την Ιταλία και την υπόλοιπη Ευρώπη, γαλλικές, ε, ντομα, γαλλικά ντοματάκια 5,70 ευρώ. 5,50 μάλλον ευρώ. Και στη Γαλλία μετά βρήκα βελγικά ντοματάκια ε, πιπεριές Ολλανδικές και όχι Ιταλικές ή Γαλλικές Ωραίες είναι οι συμφωνίες λοιπόν με τις άλλες χώρες, αλλά ίσως είναι και αναγκαίο να είμαστε κάπως λιγότερο σχεζοφρενείς στην προσέγγιση μας. Να έχουμε και λίγο πολιτικές ε, σκοπιμότητες και επιχειρήματα. Η σύνδεση με την Ουκρανία ή τη Γεωργία είναι στροφή προς, τα, προς Ανατολάς. Αλλά να ξεχνάμε ότι υπάρχει κάτι και στο νότο της Ευρώπης. Απέναντί μας υπάρχει ένας κόσμος πείνα και εξαθλίωση και ανθρώπων που δραπετεύουν για να φτάσουν στην Ευρώπη. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Δυστυχώ δεν θα έχουμε χρόνο να ακούσουμε του συναδέλφου από την ε, Γενική Διεύθυνση Άγκρη. Δεν προλαβαίνουμε. Η γνωματευσή σα υπάρχει έτσι καλώ σαν το σχέμα, οπότε απευθεία θα ακολουθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τον κύριο Τζοαν Κλάρκ. Thank you, uh, Professor Moreira. Ευχαριστώ πολύ καθηγητά Μορέρα. Λίγες σύντομες παρατηρήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις που απευθύνθηκαν στην Επιτροπή Οικονομικές Επιπτώσεις και Μηχανισμοί Ελέγχου. Ακριβώς. Οικονομικές επιπτώσεις θεωρούμε ότι θα ωφελήσει και τους εξαγωγείς της Ευρώπης και τους Μαροκινούς. Είναι κλειστή η αγορά αυτή τη στιγμή, απελευθερωμένο είναι το 1% μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ τώρα θα ανοίξει η μαροκινή αγορά και θα πάει στο 70% άνοιγμα. Ενώ ε, εμεί έχουμε μόνο το 55%. Ε, αλλά λοιπόν η μαροκινή πλευρά ή οι αναπτυσσόμενες χώρες ανοίγουν περισσότερο την αγορά από μας. Κάνουν μεγάλη προσπάθεια και πρέπει αυτό να αναγνωριστεί, να ανταμυφθεί και όχι να τιμωρηθεί. Η συμφωνία μπορεί να διορθώνει τις ανισορροπίες και το έλλειμμα που έχουμε στο γεωργικό εμπόριο με το Μαρόκο. Ε, για τις επιπτώσεις από την πλευρά της Ένωσης υπολογίζουμε ότι θα χάσουμε έσοδα από τελωνιακούς δασμούς 22 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό όμως είναι αμεληταίο. Από τη μαροκινή πλευρά υπολόγισαν ότι η νέα συμφωνία θα οδηγήσει σε απώλεια τελωνιακών δασμών, δασμών που δεν θα έχουμε να πληρώνουμε τους, για τους εξαγωγείς, 100 εκατομμυρίων. Οπότε πάλι η προσπάθεια των Μαροκινών είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δικιά μας. Επίση, γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο ευαίσθητο είναι το τομέα των οπωροκυπευτικών στην Ευρώπη, ακριβώ επειδή ξέρουμε την ευαισθησία του, επειδή πέρασε μεγάλε δυσκολίε, ακριβώ γι' αυτό αντιμετωπίσαμε μεγάλη φροντίδα στι διαπραγματεύσει στον τομέα, δεν απελευθερώσαμε τα οπωροκυπευτικά ε, διευρύναμε ε, κατά τη τις υφιστάμενες ποσοστώσεις και ε, για τις ντομάτες για παράδειγμα εκτός από ε, μία μικρή πρόσθετη ποσόστοση, η ποσόστοση αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός ε, της ε, εποχής παραγωγής στην Ευρώπη. Φθηνό, ε, όχι, χειμώνα και άνοιξη για να μην ανταγωνίζεται τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Ε, ε, Επίση, οι νέες διασφαλίσεις θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικές από τις υφιστάμενες και ακούσαμε εδώ τον κλάδο. Το σύστημα τιμών εισόδου εισαγωγή ε, το οποίο ε, το θέλουν οι εξαγωγείς μας ε, παραμένει. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν πιστεύουμε ότι η συμφωνία θα ωφελήσει τους Ευρωπαίους παραγωγούς, λαμβάνει υπόψη τι ευαισθησίε και θα ωφελήσει και το Μαρόκο. Ετέθη μια ερώτηση σχετικά με το αν θα ωφελήσει τις μικρούς αγρότες στο Μαρόκο. Αυτό δεν θα το απαντήσω εγώ, θα το απαντήσουν οι Μαροκινοί ο συνεταιρισμός λέει ναι, το 70% έχουν λιγότερο από 5 εκτάρια και 1% έχουν μόνο 50 εκτάρια. Οι συνεταιρισμοί του Μαρόκου μας έγραψαν και σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπάρχουν και αναφορές στον τύπο και λένε ότι οι μικροί που οργανώνονται σε συνεταιρισμούς τι θέλουν τη συμφωνία. Τέλος, ε, για τα θέματα SPS, ε, οι επιθεωρητές ε, για την υγεία και την ασφάλεια έκαναν και τα φυτογειονομικά έκαναν ελέγχους και έδωσαν την έγκρισή τους σε σχέση με την υγεία των προϊόντων από το Μαρόκο. Ε, και μάλιστα είναι και αυστηρά τα πρότυπα των ελέγχων αυτών. Ελπίζω να διευκρίνησα κάποια θέματα, μου είπατε να τελειώνω. Α, σε σχέση με τον εισηγητή θα υπάρξει το Μάρτιο έγγραφο εργασίας που δίνει ε, εκτενή αξιολόγηση του περιεχομένου και των επιπτώσεων της συμφωνίας και θα πρέπει να δοθεί στα μέλη του ΙΣΥΝΤ από τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει ένα εκτενές έγγραφο από την Κομισιόν που δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Οι διερμηνείς μας έδωσαν μερικά λεπτά παραπάνω, αρκετά για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ο εισηγητής έχει το λόγο. Ο κύριος Μποβέ, έχετε το λόγο κύριε Μποβέ. Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ όλους τους προσκεκλημένους μας εδώ. Ήταν σημαντικό να έχουμε ακούσει όλους τους ενδιαφερόμενους. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, άκουσα τη συζήτηση, άκουσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έμαθα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι τον Μάρτιο θα έχουμε πληροφορίες όσον αφορά τον αντίκτυπο. Αυτό σημαίνει ξεκάθαρο ότι μέχρι τώρα δεν το είχαμε και ότι αν σήμερα δεν γινόταν η συζήτηση που έγινε, δεν θα το είχαμε ούτε το Μάρτιο. Λοιπόν, είμαι επιφυλακτικό. Περιμένω να δω τι θα λέει η έκθεση αυτή του Μαρτίου. Είναι σημαντικό να την συζητήσουμε τότε και να καταλήξουμε. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειε, αλλά θα δείξω κάποια στοιχεία. Τιμή εισόδου, ευρωπαϊκές ποσοστώσει, έλεγχο στα σύνορα, όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα σε βαθμό μάλιστα που στην Επιτροπή Αναφορών υπάρχει αναφορά για αυτό το θέμα. Έπειτα το θέμα των διαφορετικών προϊόντων, εσπεροειδοειδή, μανταρίνια, ντομάτα, υπάρχει στρέβλωση τιμών και εδώ χρειάζεται συζήτηση. Έπειτα το θέμα των ποσοστώσεων το αναφέραμε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τρεις επιχειρήσεις οι οποίες τελικά ελέγχουν πάνω από το 70% των εξαγωγών από το Μαρόκο, δύο ευρωπαϊκών κεφαλαίων, γαλλικών. Εμένα μου φαίνεται αυτό ότι έρχεται σε αντίφαση με τα όσα Ακούσαμε ότι είναι υπέρ της ανάπτυξης των μικρών παραγωγών του Μαρόκου. Κάτι άλλο, σήμερα ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές γές που δίνονται σε ξένες επιχειρήσεις, σε κονσόρσια μάλιστα, τα οποία φτιάχνονται στο Μαρόκο, σε βάρος βέβαια των τόπιων. Και υπάρχει κριτική και μέσα στο Μαρόκο από γεωπόνους μαροκινούς οι οποίοι λένε ότι αυτά τα σχέδια είναι σε βάρος της πλειοψηφίας των Μαροκινών γεωργών. Τρία ακόμα σημαντικά σημεία. Όχι με λεπτομέρειες. Το δικαίωμα ε, εργασίας, το εργασιακό δίκαιο. Τα συνδικάτα διαμαρτύρονται. Υπάρχουν ε, όμως τα δικαιώματα των ε, μισθωτών γεωργών, τα οποία παραβιάζονται, ενώ αναγνωρίζονται κανονικά διεθνώ όσον αφορά τι εξαγωγέ αυτέ προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το νερό και τη χρήση του, δεν χρειάζεται να πω περισσότερο, το θέμα του νερού εννοείται ότι είναι κεντρική σημασία, διότι σήμερα οι εξαγωγέ που έρχονται από το Μαρόκο αντιστοιχούν σε 25 εκατομμύρια κυβικά νερού. Δηλαδή σήμερα εξάγουν προς την Ευρώπη 25 εκατομμύρια κυβικά από μια χώρα δηλαδή η οποία υποφέρει και έχει προβλήματα στον υδροφόρο της ε, ορίζοντα από έλλειψη νερού και που δεν έχουν και άλλους σπόρους. Τέλος, το περιμένατε, το θέμα της διοικητικής εντό αγωγικών δύναμης της Δυτικής Σαχάρας. Αναφερθήκαμε και σε αυτό, αλλά τι διαπιστώνουμε. Διαπιστώνουμε ότι οι εξαγωγείς όπως η Αζούρα, η, η έχουν εκεί τη βάση τους και το κάνουν σε βάρος του ντόπιου πληθυσμού. Αν δούμε την νομική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα, διαπιστώνουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να πει κατά πόσο συμφωνία αυτή συνάδει με το διεθνές δίκαιο. Όταν βλέπουμε τι απάντηση έδωσε η Επιτροπή του κύριου Παρόσο για να μας πει ότι σέβεται τις συμφωνίες, εγώ λέω ότι δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για να το πούμε αυτό. Συνεπώς σήμερα ζητάω ξεκάθαρα στο όνομα, τελειώνω, τελειώνω πρόεδρε, στο όνομα λοιπόν του άρθρου 90 σημείο 6 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 268 ενδέκατη παύλα του ε, κειμένου ίδρυσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ζητάω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορίου Επιτροπή μας ε, δηλαδή να υποβάλει αίτημα στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου μας, ώστε το Κοινοβούλιο να θέσει αίτημα κατά πόσο συνάδει η συμφωνία αυτή με το Διεθνές Δίκαιο και να απευθυνθεί γι' αυτό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οπότε ζητάω από τον πρόεδρο της Επιτροπής μας, Ίντα, να μεταφέρει στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το αίτημα αυτό βάσει, όπως σας είπα, του άρθρου 90 του κανονισμού σημείο 6. Είναι, πιστεύω, κάτι πολύ σημαντικό αν θέλουμε οριστικά να λύσουμε το θέμα του κατά πόσο όλα αυτά συμμορφώνονται στο Εθνές Δίκαιο ή όχι. Μάλιστα, το λαμβάνω υπόψη μου λέει ο πρόεδρος. Εγώ έχω το λόγο, λέει ο πρόεδρος. Είναι οι ευρωβουλευτές που αποφασίζουν γι' αυτό, όχι εγώ. Για το χρονοδιάγραμμα τώρα. Ο εισηγητής προτείνει το εξής χρονοδιάγραμμα. Σχέδιο έκθεσης. 12 Οκτωβρίου να είναι έτοιμο, να σταλεί στη μετάφραση, να μπορέσουμε να το εξετάσουμε στις 22 Νοεμβρίου στην Επιτροπή μας. Προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών 25 Νοεμβρίου. Θα ψηφίσουμε το Δεκέμβριο στην Επιτροπή μας. και θα πάει στις 20 Δεκεμβρίου και θα πάει στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο. Εντάξει, συμφωνείτε με το χρονοδιάγραμμα. Κύριε Μποβέ, έχω αντίρρηση, λέει ο κύριο Μποβέ. Δεν μπορούμε σήμερα. Εγώ επίσημα σας υπέβαλα ένα αίτημα εφαρμογής του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν μπορείτε να παρακάμψετε αυτή την υποχρέωση. Μα δεν είναι δικό μου θέμα, λέει ο Πρόεδρος. Εγώ απορρίπτω το αίτημά σας και το χρονοδιάγραμμα το οποίο εσείς έχετε προτείνει ως εισηγητής, αυτό θέτω σε ψηφοφορία να μας πούνε τα μέλη των συμφωνούν. Δεν μπορείτε τώρα να έρχεστε τελευταία στιγμή έτσι να προσπαθείτε να αναβάλλετε για άλλη μια φορά αυτή την υπόθεση. Το χρονοδιάγραμμα εσείς ο ίδιος το έχετε προτείνει. Το έτομά σα δεν είναι για μένα, δεν εξαρτάται από μένα ούτε καν από την Επιτροπή μας. Οπότε θέτω σε ψηφοφορία το σχέδιο χρονοδιάγραμματος που εσείς ο ίδιος προτείνετε στην Επιτροπή μας. Πρέπει να είστε συνεπείς, Μποβέ. Διακόπτει ο κύριος Μποβέ. Πρόεδρε, προσπαθώ να χρησιμοποιήσω το δικαίωμά μου. Σας διαβάζω στα γαλλικά για να είναι ξεκάθαρο. Τι λέει εδώ, λέει ο κανονισμός ότι πριν τεθεί σε ψηφοφορία, πρόεδρος τον διακόπτη. Μιλάνε μαζί. Το άκουσα το έτοιμά σας. Αυτό που σας λέω κύριε Μποβέ είναι ότι δεν εξαρτάται από μένα να αποφασίσω. Οπότε ψηφίζουμε το χρονοδιάγραμμα που προτείνατε εσείς ο ίδιος. Αυτό προτείνω στην Επιτροπή μας. Πρόεδρε Διακόπτη, κύριε Σποβέ, τα είπατε, ό,τι είχατε να πείτε το είπατε. Παραβιάζετε τον κανονισμό Ρωτήστε τις ε, νομικές υπηρεσίε να σα το επιβεβαιώσουν, λέει ο κύριο Βοβέ. Διακόπτε ο πρόεδρος, άκουσα το έτοιμά σα. Εγώ απέρριψα το έτοιμά σα και ψηφίζουμε το χρονοδιάγραμμα. Όχι, λέει ο κύριο Μποβέ, δεν συμφωνούμε. Με εδώ υπάρχει ένα συμβιβασμό. Εγώ δέχτηκα την πρότασή σας αλλά υπό τον όρο ότι δεν θα προσπαθούσατε να αναβάλλετε πάπυρο αυτή την υπόθεση. Αυτή ήταν μια συμφωνία κυρίων που είχαμε κάνει δυο μας, εσείς με μένα. Τώρα παραβιάζετε αυτή τη συμφωνία. Δεν πρόκειται μόνο για θέμα ε, νομικών προδιαγραφών, πρόκειται για συμφωνία κυρίων. Κάνατε μια τέτοια συμφωνία μαζί μου και τώρα την παραβιάζετε. Μποβέ, μα υπάρχει δίκαιο, εδώ δεν κάνουμε σχόλια. Το δίκαιο το αποφασίζω εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Ψηφίζουμε το χρονοδιάγραμμα. Μα υπάρχουν κείμενα. Βάσει των κειμένων έχουμε το δίκαιο. Πρόεδρος, είπατε ότι είχατε να πείτε. Ψηφίζουμε το χρονοδιάγραμμα. Ποιο είναι υπέρ του χρονοδιαγράμματος έτσι όπως αυτό προτείνεται από τον εισηγητή. Ποιος συμφωνεί με το χρονοδιάγραμμα αυτό που έχει προτείνει ο εισηγητής, ο πρόεδρο. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Εγκρίνεται. And we'll move to the conclusion of this... Uh, Και έτσι ολοκληρώνεται η συνεδρίαση αυτή. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Έληξε συνεδρίαση.